Μπορούμε να ξεκινήσουμε τις εργασίες μας σήμερα το απόγευμα. Ήδη δουλέψαμε καλά νομίζω το πρωί, αντιμετωπίζοντας το θέμα του ενιαίου εκλογικού συστήματος. Τώρα θα πρέπει από κοινού να περάσουμε στην συζήτηση με τα κοινοβούλια των κρατών μελών για την πρωτοβουλία των πολιτών. Το θέμα αυτό θα παρουσιαστεί από τους τέσσερις εισηγητές. Έχουμε δύο εισηγητές για την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων και δύο για την Επιτροπή των Αναφορών. Γκουρμάι, Λαμασούρ, Έφνερ και Βόλις για την Επιτροπή Αναφορών. Όπως βλέπετε όλες περίπου οι πολιτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εκπροσωπούνται μέσω αυτών των τεσσάρων επιτρόπων και αυτό νομίζω ότι δείχνει το βάρος που δίνουμε στο συγκεκριμένο θέμα. Ο πρόεδρος Φλαό δεν μπόρεσε να πάρει μέρος στη συνάντησή μας και αντικαθίσταται από την κυρία Ρούτεν, την οποία θα ήθελα να χαιρετήσω. Και έχουμε εδώ και τον κύριο Σαστέλ. Ήταν α, ε, επίσης ε, γνωστός μας. Έχουμε και τον κύριο Σεύκοβιτς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον Επίτροπο Σεύκοβιτς. Και γι' αυτό θα ήθελα παρακαλώ όπως κάναμε και το πρωί αυτοί οι οποίοι θα ήθελαν το λόγο να συμπληρώσουν το δελτίο το οποίο έχουν στη διάθεσή τους έτσι ώστε να μπορέσουμε να οργανώσουμε σωστά την συζήτηση. Πριν από δώσω το λόγο στους τέσσερις ομιλητές, θα ήθελα να πω ότι με τις εργασίες μας συνδέεται σήμερα η Επιτροπή Φυσικά Αναφορών και αυτό αποδεικνύεται από την παρουσία και των δύο εισηγητών και φυσικά από την πρόεδρο της Επιτροπής θα έρθει ο πρόεδρος σε λίγη ώρα και θα συμπροεδρεύσει. Θα ήθελα να ζητήσω τώρα από την κυρία Ρούτεν να κάνει τον αρχικό χαιρετισμό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Σαν βουλευτής της Βελγικής Βουλής και σαν τέος υπάλληλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι τιμή μου να πάρω μέρος σήμερα ε, στην συνεδρίαση αυτή της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων με προσκεκλημένα τα κοινοβούλια των κρατών μελών. Ο Αντρέ ο πρόοδος της Βουλής, είναι διαμεσολαβητής για τον σχηματισμό της νέας βελγικής κυβέρνησης και αδυνατή να πάρει μέρος στη συνάντησή σας σήμερα. Θα ήθελα να, του να σας μεταφέρω το μήνυμά του μετά από τις προσπάθειες που έγιναν κατά τη διάρκεια των προηγούμενων προεδριών του Συμβουλίου, η Βελγική Προεδρία έχει αποφασίσει να βοηθήσει έτσι ώστε οι διαδικασίες μετά από τη συνθήκη της Λισαβόνας να γίνουν ακόμα πιο διαφανείς η Βελγική Προεδρία θα προσπαθήσει να κάνει γνωστή την Ευρωπαϊκή Ένωση στον υπόλοιπο κόσμο αλλά και στο εσωτερικό της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή στους πολίτες της. Ένας από τους στόχους για να το πετύχουμε αυτό είναι η πρωτοβουλία των πολιτών. Είναι μια βασική καινοτομία της συνθήκης της Λισαβόνας. Ήδη από το 1979 μπόρεσαν οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να πάρουν μέρος ε, με καθολική ψηφοφορία στην εκλογή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τώρα πλέον μέσω της συνθήκης της Λισαβόνας τους δίδεται η δυνατότητα να ακουστεί η φωνή τους άμεσα και αυτό είναι βασικό ε, σημείο πρόοδου. Όπως γνωρίζετε πολύ καλά η αρχή της λαϊκής πρωτοβουλίας εγγράφεται στο άρθρο 11 σημείο 4 της συνθήκης που λέγει ότι ε, ένα τουλάχιστον εκατομμύριο πολιτών της Ευρώπης από ένα σημαντικό αριθμό κρατών μπορούν να πάρουν την πρωτοβουλία να προσκαλέσουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταθέσει μια κατάλληλη πρόταση στο θέμα στο οποίο θεωρούν οι πολίτες ότι μια δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι απαραίτητη στα πλαίσια της εφαρμογής της συνθήκης. Η συνθήκη της Λισαβόνας λοιπόν έχει ξεκινήσει το δρόμο στη συμμετοχική δημοκρατία η μέθοδος αυτή συμπληρώνει την αντιπροσωπευτική δημοκρατία στην οποία εδράζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Καθιερώνεται επίσης και η υπάρχουσα πρακτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ξεκινά δημόσιες διαβουλεύσεις έτσι ώστε να δοθεί δυνατότητα στους πολίτες να γνωστοποιήσουν την άποψή τους πριν προχωρήσει στην πρόταση ε, νομοθετική, ε, νομοθετικής, ε, νομοθετικού περιεχομένου. Τα θέματα των διαδικασιών για τη λειτουργία αυτού του, αυτής της μεθόδου θα πρέπει να συζητηθούν έτσι περαιτέρω στα πλαίσια του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου. Η Βελγική Προεδρία θέλει να πάρει μέρος στην προώθηση αυτού του καινοτόμου προγράμματος ε, διαθέτοντας ε, ε, χρόνο και τεχνολογικά μέσα. Η μέθοδος αυτή όχι μόνο θα μπορέσει Ζητώ συγγνώμη λέει η ομιλήτρια γιατί διαβάζω πολύ γρήγορα. Θέλουμε να δημιουργήσουμε μια γέφυρα ανάμεσα στο παρόν και το παρελθόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι τεχνολογίες ε, της επικοινωνίας ανήκουν πλέον ε, στην καθημερινότητά μας και μέσω του παγκοσμίου διαδικτύου τα φόρουμ πολλαπλασιάζονται συνεχώς. Το σχέδιο λοιπόν αυτό λαϊκής πρωτοβουλίας νομίζω ανοίγει νέε δυνατότητες επιτρέποντας την έκφραση ε, των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ηλεκτρονική ε, μορφή αυτής της ε, διαδικασίας νομίζω ότι πρέπει να μας καταστήσει ιδιαίτερα προσεκτικούς γιατί θα πρέπει εμείς τις διαδικασίες να τις κρατήσουμε απλές και ελεγχόμενες χωρίς να επιβαρύνουμε γραφειοκρατικά τις υπηρεσίες των κρατών μελών, διασφαλίζοντας την ασφάλεια του συστήματος και τις πιθανές καταχρήσεις. Νομίζω ότι έχουμε αρκετές δυνατότητες και η προοπτική αυτή μπορεί στην ουσία να οδηγήσει στην αναγέννηση της ιδέας της άμεσης δημοκρατίας όπως ασκήθηκε στην αρχαία αγορά της αθηναϊκής δημοκρατίας Νομίζουμε ότι στην ουσία έχουμε να κάνουμε με την αναγέννηση μιας πολιτικής μεθόδου η οποία προέρχεται από μια σημερινή χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης την οποία ονομάζουμε πολύ συχνά η κοιτίδα της δημοκρατίας. Πάντως μένει πολλά να γίνουν ακόμα και ελπίζουμε η δημοκρατική συμμετοχή στην προσπάθεια της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης θα ενισχυθεί ακόμα περισσότερο. Πέρα από αυτόν τον πρώτο στόχο, καλό θα είναι να προσπαθήσουμε το κοινοτικό αυτό μέσο να προχωρήσει, να επιτρέψει στην ενίσχυση του ευρωπαϊκού χώρου και να ευνοήσει την κοινωνική συνοχή, συμμετέχοντας στην διαμόρφωση μιας ευρωπαϊκής πλέον και όχι εθνικών κοινή γνώμης. Μία προσωπική παρατήρηση η πρωτοβουλία των πολιτών είναι μια εξαιρετική επίσης ευκαιρία να φτάσουμε κοντά στους νέους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να παραμένει ένα σχέδιο για το μέλλον και να προωθεί την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση ανάμεσα στους νέους της Ευρώπης. Αυτός θα πρέπει να είναι ο κεντρικός μας στόχος. Είμαι πεπισμένος ότι ε, ε, σε αυτό θα βοηθήσει επίσης και η δυνατότητα να ψηφίζουν οι νέοι στις ευρωεκλογέ από την ηλικία των 16 ετών. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και ε, εκ μέρους του κυρίου Φλαό σας εύχομαι καλή τύχη στις εργασίες σας. Ευχαριστούμε πολύ. Ε, στο σημείο αυτό ε, προβλέπεται στο πρόγραμμα η παρέμβαση της κυρίας Ματσόνη ε, που είναι πρόεδρος της Συνδεδεμένης Επιτροπής. Αλλά εφόσον δεν είναι εδώ η κυρία Ματσόνη πώς να την ακούσουμε. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να επενθυμίσω το εξή, ότι πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία, αυτή η πρωτοβουλία των πολιτών. Αυτό ήδη ελέγχθη το άρθρο 11 τέταρτο κόμμα της ε, Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση της Συνθήκης της Λισαβόνας προβλέπει τη θέσπιση αυτής της ε, πρωτοβουλίας των πολιτών. Όμως, εναπόκειται σε εμά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να καταθέσουμε ένα σχέδιο το οποίο θα περιλαμβάνει επακριβώς τους κανονισμούς που θα διέπουν αυτή την καινοτομία. Έχουμε ε, προχωρήσει στη δουλειά μας και στις 8 Νοεμβρίου προβλέπεται οι εισηγητές να καταθέσουν τη δική τους την πρόταση προς την Επιτροπή. Γι' αυτό λοιπόν αυτή η συνεδρίαση έχει πολύ μεγάλη σημασία για να κατατεθούν και ενδεχομένω τροπολογίε και για να αξιολογηθεί η μέχρι τώρα εργασία. Τη μεγαλύτερη δουλειά την έχουν οι συγητέ. Θα ακούσουμε λοιπόν τους συγητές και μετά θα ακούσουμε και τους ε, αρμόδιους από το Συμβουλίο και από την ε, Επιτροπή. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο για πέντε λεπτά, όχι παραπάνω, στους εισηγητές. Δεν ξέρω ποιος θέλει να ξεκινήσει. Ίσως ο πρόεδρος κύριος Λαμασούρ. Κύριε Λαμασούρ, ε, θέλετε να ξεκινήσετε, να μας πείτε τη δική σας άποψη. Παρακαλώ. Je voudrais, euh, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ξεκινήσω υπενθυμίζοντάς σας πώς ξεκίνησε από τη συνθήκη της Λισαβόνας βέβαια, όπως πολύ σωστά είπε ο Πρόεδρος, που προβλέπει την πρωτοβουλία αυτή ως δικαίωμα των πολιτών. Υπήρξαν πολλές διαδικασίες, χαιρετίζω και τον Επίτροπο Σπάκοβιτς εδώ πέρα, και έτσι πριν ξεκινήσει οποιαδήποτε νομοθετική πρωτοβουλία, φροντίζει η Επιτροπή να έρθει σε διαβούλευση όχι μόνο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με τα Εθνικά Κοινοβούλια, με τις κυβερνήσεις, αλλά και με τους κοινωνικούς εταίρους, τα συνδικάτα, τις μη κυβερνητικές οργανώσεις κλπ. κλπ μέσω δημοσίευσης μιας πράσινης βίβλου, μια λευκής βίβλου κλπ. Έπειτα, το ίδιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, επιμονή μου βάσεως, οργανώνει φόρα με ανταλλαγές εμπειριών, πληροφοριών, συζητήσεις με την ΟΚΕ, με την Επιτροπή των Περιφερειών και η Επιτροπή Αναφορών, η δικιά μας, οι συγητές από την Επιτροπή αυτή θα το πούν, φροντίζει για τις επαφές αυτές με τους Ευρωπαίους πολίτες. Όμως έχουμε μεγάλα προβλήματα. Το ένα μεγάλο πρόβλημα που είναι ένα μόνιμο πρόβλημα που έχουμε και με το οποίο πρέπει να μάθουμε να ζούμε είναι ότι οι Βρυξέλλες είναι μακριά από τον πολίτη. Και όπως λοιπόν οι εθνικές μας πρωτεύουσες είναι μακριά από τους πολίτες, σε αναλογία με το που βρίσκονται οι πρωτεύουσες των περιφερειών, εννοείται ότι πάντα οι Βρυξέλλες θα είναι μακριά από τις πρωτεύουσες των χωρών. Έτσι λοιπόν, σε αντίθεση με το τι ισχύει στα ομοσπονδιακά συστήματα, δεν υπάρχει ευρωπαϊκή δίκηση εκτός Βρυξελών. Δεν υπάρχει δηλαδή ευρωπαϊκή γραφειοκρατία. Δηλαδή όλοι οι υπάλληλοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι στις Βρυξέλλες, μακριά από τις χώρες. Και το κοινοτικό δίκαιο τίθεται σε εφαρμογή από τις εθνικές και περιφερειακές αρχές και οι πληροφορίες για το κοινοτικό δίκαιο δίνονται από τις εθνικές και περιφερειακές αρχές στον κόσμο. Το άλλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε και για το οποίο πρέπει να βρούμε λύση είναι ότι όλος παραδόξως μετά από 50 χρόνια οικοδόμησης της Ευρώπης, 50 χρόνια κατά διάρκεια των οποίων καταργήσαμε ε, τους φραγμούς μεταξύ μας, τα σύνορα, τους ελέγχους στα σύνορα. Η κυκλοφορία είναι ελεύθερη για τους πολίτες, για τα εμπορεύματα, για τα γεωργικά προϊόντα, για τις πληροφορίες, για τα κεφάλαια. Όμως όχι για την πολιτική συζήτηση. Εξακολουθούμε να ζούμε μέσα σε 27 διαφορετικές πολιτικές συζητήσεις που γίνονται ξεχωριστά στην κάθε μία από τις χώρες μας. Και με τις εκλογές κάθε πέντε χρόνια είναι λίγο πολύ 27 διαφορετικές εθνικές εκλογές με ένα πρόσχημα ευρωπαϊκό. Δεν είναι πραγματικά ευρωπαϊκή συζήτηση που γίνεται για τις εκλογές αυτές. Παράδειγμα στη Γαλλία, στη χώρα μου. Η, το κύριο κανάλι πληροφόρησης, η TF1, της τηλεόρασης, που ένα τρίτο των Γάλλων στις 20 κοιτάνε τις ειδήσει κάθε βράδυ, δεν έχει μόνιμο ανταποκριτή στις Βρυξέλλες. Αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι η γαλλική τηλεόραση μιλάει για την ευρωπαϊκή ζωή μόνο αν κάποιος από τις γαλλικές αρχές έρθει στις Βρυξέλλες. Και τότε έρχονται και οι δημοσιογράφοι, τραβάνε εικόνες και τότε παρουσιάζουν μια καθαρά εθνική οπτική γωνία της ευρωπαϊκής πολιτικής στους Γάλλους πολίτες. Και φοβάμαι ότι και στις άλλες χώρες το ίδιο γίνεται. Εξού και ιδέα αυτής της διαδικασίας είναι μια πρωτότυπη διαδικασία η οποία δεν υπάρχει στις χώρες μας. Ε, σε κάποιες χώρες υπάρχει κάτι που μοιάζει. Δεν είναι αναφορά, όπως την ξέρουμε, και δεν είναι δημοψήφισμα, δεν είναι απευθείας ε, δημοκρατία καθολική, τι προσπαθούμε εμεί να κάνουμε με την πρωτοβουλία αυτή. Προσπαθούμε να δώσουμε στον Ευρωπαίο πολίτη, στους Ευρωπαίους πολίτες, εφόσον είναι αρκετοί, ένα εκατομμύριο και προέρχονται από πολλέ διαφορετικές χώρες, θέλουμε λοιπόν να τους δώσουμε το ίδιο, την ίδια ισχύ, την ίδια εξουσία να μπορούν να βάλουν μπρο για μια ε, πολιτική και νομική διευθέτηση όπως μπορεί σήμερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο Υπουργών. Σήμερα τα νομοθετικά σώματα είναι το Συμβούλιο των Υπουργών και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μπορούν όμως να αναλάβουν και πολιτικές πρωτοβουλίες. Αυτές οι πολιτικές πρωτοβουλίες καταλήγουν σε νομοθεσία εφόσον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το αποφασίσει. Είναι αυτό δηλαδή η κύρια ευθύνη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν μπορούμε δηλαδή να φτιάξουμε νόμους αν δεν έχουμε προηγουμένως κάποια γραπτή πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό είναι το λεγόμενο μονοπόλιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι ένα νομικό ε, μονοπόλιο, αλλά δεν έχει και το μονοπόλιο των πολιτικών ιδεών. Και η εμπειρία έχει δείξει, το βλέπουμε από τα στατιστικά δεδομένα που έχουμε, ότι σε 10-15 χρόνια, τα τελευταία δηλαδή 10-15 χρόνια, οι πολιτικές πρωτοβουλίες για νέες πολιτικές ή για νέα νομοθεσία, λίγο πολύ μοιράζεται ένα τρίτο, ένα τρίτο, ένα τρίτο, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Τι, τι προτείνουμε εμείς λοιπόν τώρα μέσα από τη συνθήκη της Λισαβόνας, προτείνουμε έναν τέταρτο αρμόδιο για να αναλάβει πολιτικές πρωτοβουλίες και αυτός είναι ο Ευρωπαίος πολίτης. Εφόσον λοιπόν αρκετοί Ευρωπαίοι πολίτες μαζευτούν μαζί, μπορούν να ζητήσουν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπό την ευθύνη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να αναλύσει την πρότασή τους και να αποφασίσει ελεύθερα, βάσει των αρμοδιοτήτων της, κατά πόσο θα δώσει συνέχεια με νομοθετική διάταξη ή μετροποποίηση τροποποίηση κάποιας νομοθετικής που ήδη υπάρχει ή όχι στην πρωτοβουλία αυτή των πολιτών. Άπαξ και διατυπώ στην πρότασή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μετά είναι στα χέρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου να συμφωνήσουν ή όχι. Τι διαδικασία προβλέπουμε τώρα, έχοντας συνεργαστεί και με τον Επίτροπο και με τον ε, Πρόεδρο η διαφορά ανάμεσα στην αναφορά και την πρωτοβουλία Ευρωπαίων πολιτών. Η αναφορά... Να, χτες είδαμε τι έγινε στους δρόμους των Βρυξελών. Είναι μια διαδικασία με την οποία ο πολίτης αναλαμβάνει ενεργά το ρόλο του. Μπορεί να ζητήσει να σταματήσει μια πρωτοβουλία ευρωπαϊκή ή ένα νόμο αυτό γίνεται με τις διαδηλώσεις. Ενώ εδώ πρόκειται για τον άποδο, πρόκειται για την θετική προσέγγιση. Άρα λοιπόν, όποιος θέλει, είτε πολιτικές ε, οργανώσεις, κόμματα, συνδικάτα κτλ. Ο κύριος στόχος όμως είναι οι Ευρωπαίοι πολίτες με τους οποίους, για τους οποίους δεν ενδιαφερόμαστε εμείς, οι πολιτικοί, είτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε από τις χώρες μας, είτε επειδή γεωγραφικά είναι διάσπαρτοι στην Ευρώπη, είτε επειδή δεν είναι αρκετά οργανωμένοι για να κάνουν τη φωνή τους να ακουστεί. Είναι Ευρωπαίοι πολίτες λοιπόν, επίσης, οι οποίοι ε, ζουν σε διαφορετική χώρα από εκείνη από την οποία έχουν ε, μεγαλώσει. Ε, παντρεύονται, κάνουν παιδιά, οικογένεια, δουλεύουν, αρρωσταίνουν, βγαίνουν στην ανεργία κλπ. Σύμφωνα με τους νόμους που εμείς ψηφίζουμε εδώ, θα έπρεπε και αυτοί να συμπεριλαμβάνονται και πολύ εύκολα να λύνονται και τα δικά τους τα προβλήματα. Όμως δεν συμβαίνει αυτό. Και έτσι πρέπει να τους δίνεται η ευκαιρία να φτάνουν ως εμάς, διαμαρτυρώμενοι, είτε ζητώντας κάτι, όχι συστηματικά για να καταστρέφουν αυτό που κάνουμε, αλλά να μπορούν να μας εξηγήσουν ποια είναι τα καθημερινά τους προβλήματα και πώς μπορούμε μαζί τους να φτιάξουμε την ομοθεσία την οποία χρειάζονται οι Ευρωπαίοι πολίτες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Λαμασούρ γιατί μας παρουσιάσατε ένα σαφέστατο πλαίσιο ιδιαίτερα πολιτιστικού θα έλεγα χαρακτήρα και θα ήθελα να ζητήσω τώρα από την κυρία Γκουρμάη την αντιπρόεδρό μας να συμπληρώσει κατά κάποιο τρόπο αυτά που είπε ο κύριος Λαμασούρ. Είναι σημαντικό το θέμα αυτό και γι' αυτό ακριβώς υπάρχουν και τέσσερις ε, ουσιαστικά εισηγητές. Το θέμα είναι όπως είπα πολύ σοβαρό και προκαλεί τεράστιο ενδιαφέρον η προσπάθεια να προχωρήσουμε σε μια κάποια ασυνένεση. Άλλωστε και η παρουσία εδώ του Σαστέλ και του Σεύκοβιτς δείχνει το μεγάλη σημασία. Και χαίρομαι που έχω πίσω μου εδώ τον κύριο Ροτ και τους άλλους εκπροσώπους από τα κοινοβούλια των κρατών μελών. Θυμίζω ότι είχαμε επίσης συζητήσεις μέχρι τώρα για το θέμα αυτό και με την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή θα έχουμε τελικά ένα καλό μέσο για την προώθηση της δημοκρατίας. Ένας μεγάλος πρόεδρος βέβαια όπως κύριος Καζίνη έχει συνεισφέρει και αυτός προς την κατεύθυνση αυτή. Θα ήθελα να σας αναφέρω λίγο το τι έχει συμβεί μέχρι τώρα. Η αλήθεια είναι ότι όπου έχει κάνει μια επιτυχημένη προσπάθεια ένας άνδρας πίσω του κρύβεται μια γυναίκα και το αντίστροφο συμβαίνει βέβαια. Ε, φαίνεται ότι κάποιοι κρύβονται πίσω από την πλάτη μου. Εν πάση περιπτώσει θα ήθελα να ευχαριστήσω όσους προώθησαν το πράσινο βιβλίο. Θα θέλαμε και κατά τη διάρκεια της Ουγγρικής Προεδρίας και είμαι ιδιαίτερα υπερήφανη που είμαι Ουγγαρέζα και οι Ούγγροι και με τους Ισπανούς θα μπορέσουν μέχρι τις 22 Ιουνίου να μας κάνουν μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση. Και έτσι και ο Μάρις και ο Σαστέλ θα συνεισφέρουν με τον δικό τους τρόπο. Θυμίζω ότι μέχρι τώρα είχαμε πάρα πολλές διαβουλεύσεις με την κοινωνία των πολιτών και όχι μόνο με όργανα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα πλαίσια μιας διαδικασίας η οποία είναι αρκετά περίπλοκη και αυτό το δείχνει και η συζήτηση που έγινε σήμερα το πρωί ε, γύρω από την πρόταση του κυρίου Νταφ. Ξέρετε ότι ε, πολλοί είναι κατά γενικά των προτάσεων οι οποίες έχουν σαν στόχο την προώθηση της ευρωπαϊκής δημοκρατίας και αυτό δυσκολεύει τα πράγματα. Πιστεύω λοιπόν ότι έχουμε και ένα σκληρό χρονοδιάγραμμα πέρα από τις δυσκολίες της ουσίας και ελπίζω θα πρέπει να γίνει μετάφραση σε όλες τις γλώσσες έτσι ώστε όλοι να έχουν ισότιμη πρόταση θα πρέπει να περιμένουμε και την γνωμοδότηση της Επιτροπής Δημοσίων Ελευθεριών όπως επίσης και τη γνωμοδότηση το, της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων. Και φυσικά ε, υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι συνεργάζονται με τον Μάρε Σεύκοβιτς και περιμένουμε από όλου να κάνουν τις προτάσεις τους τώρα που έχει προχωρήσει σχετικά η διαδικασία. Ο χρόνος είναι πλέον καλός για να γίνουν συζητήσεις με τα κοινοβούλια των κρατών μελών. Σήμερα το πρωί υπήρξαν 26 σχόλια στην έκθεση του ΝΤΑΦ. Ελπίζω να προκληθεί το ίδιο ενδιαφέρον και για τις προτάσεις οι οποίες γίνονται σήμερα το απόγευμα. Προφανώς θα θέλαμε να βελτιώσουμε την πρόταση του ψηφίσματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εμείς θέλουμε να καταστήσουμε πιο φιλικό στο χρήστη ε, το συγκεκριμένο σύστημα, την συγκεκριμένη μέθοδο. Πρόκειται για ένα ισχυρότατο δημοκρατικό μέσο. Δεν θα πρέπει να υφίσταται κατά χρήση, θα πρέπει να λειτουργεί με χρήσιμο τρόπο. Γίνονται βέβαια κάποιες συζητήσεις για το πότε θα ξεκινήσουμε το 2016 ή κάποια άλλη στιγμή. Η Ευρώπη είναι ανοιχτή σε όλους και ας ελπίσουμε ότι τα κράτη-μέλη είναι διατεθειμένα να βοηθήσουν και να αλλάξουν τις νομοθετικές ρυθμίσεις. Θα κάνουμε κάποιες προτάσεις στην πρόταση ψηφίσματος έτσι ώστε να αποφύγουμε γραφειοκρατικές καθυστερήσεις. Να σας δώσω ένα παράδειγμα του τι μπορούμε να κάνουμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέγει ότι θα ελέγχει το αποδεκτό κάποιων τέτοιων λαϊκών πρωτοβουλειών εφόσον συμπληρωθεί ο αριθμός των 300.000 υπογραφών. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να συζητήσουμε για να μην δημιουργηθούν παρανοήσεις. Το θέμα είναι τι θα γίνει και στο τέλος της διαδικασίας. Όταν συγκεντρωθούν σαν παράδειγμα όλες αυτές οι υπογραφές, τι θα γίνει θα πρέπει να υπάρξει μια κάποια ανταπόδοση θα έλεγα, ένα κάποιο μήνυμα, μια ακρόαση για να συνεχιστεί η επαφή ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους πολίτες. Ο κύριος Λαμασούρ θα δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά έχει σημασία ο τρόπος που θα λειτουργήσει η διαδικασία αυτή. Προσπαθούμε εμείς να καθορίσουμε τη διαδικασία στη λεπτομέρειά της και να την καταστήσουμε χρησιμοποιήσιμη το ταχύτερο δυνατόν μέχρι το τέλος του χρόνου, σαν δώρο γενεθλίων θα έλεγα για τη συνθήκη της Λισαβόνας. Νομίζω ότι έχουμε κάποιο χρόνο έτσι ώστε να μπορέσουμε να προωθήσουμε ε, την προσπάθεια αυτή προς το καλό των πολιτών. Με αυτό το στόχο είμαστε πάντα διατεθειμένοι για τις προτάσεις όλων σας εδώ και από τα κοινοβούλια των κρατών μελών και από τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που επιδεικνύουν ισχυρότατο ενδιαφέρον Ας τα έχετε όλα αυτά υπόψη σας λοιπόν, εμείς σας μην επιβραδύνουμε την διαδικασία αυτή, χωρίς όμως να επιτρέψουμε την υψηλή ταχύτητα αυτής της διαδικασίας να χαμηλώσει την ποιότητά της. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Γκουρμάη. Ε, δεν ξέρω ποιος θέλει να μιλήσει. Κυρία Γουόλης παρακαλώ. Πρόεδρε, επειδή ε, νομίζω ότι ε, τώρα πια έχουν έρθει όλοι στην αίθουσα, ο Στερχόντσεν, είναι μια ομαδική εργασία ανάμεσα στους εισηγητές, ε, τους θεσμούς και θα πρέπει αυτή η ομαδική εργασία να επεκταθεί και στα εθνικά κοινοβούλια γιατί δεν θα μπορέσουμε ποτέ να πετύχουμε τον Ευρωπαϊκό Δημοκρατικό Χώρο, για τον οποίο έγινε επανειλημμένα λόγος, αν δεν συνεργαστούμε με τους εθνικούς συναδέλφους στα κράτη-μέλη. Εκείνο λοιπόν που θέλουμε να συστήσουμε εδώ είναι κάτι το οποίο να είναι ελκυστικό και προσπελάσιμο για τους πολίτες. Πάνω απ' όλα το δεύτερο. Άρα δηλαδή οφείλουμε να συμμετέχουμε στην ευρωπαϊκή ε, δημοκρατία. Εξετάζω αυτό το θέμα ο συνάδελφός μου από την ε, Επιτροπή Αναφορών και άλλοι εμπνεύστηκαν από την εμπειρία που συγκεντρώθηκε ε, όλα αυτά τα χρόνια από το δικαίωμα των Εβραίων πολιτών να καταφεύγουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό δικαίωμα, το δικαίωμα προσφυγής. Ε, το έχουν όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες. Και έτσι λοιπόν βλέπουμε πώς ε, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μία διαδικασία. Θα πρέπει να είναι σαφές ότι η ευρωπαϊκή διαδικασία κατάθεσης αναφορών δεν είναι ακριβώς το ίδιο όπως και οι δυνατότητε συμμετοχή, όμως είναι χρήσιμη αυτή η εμπειρία. Και ε, θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο πράγματα. Ε, το δικαίωμα ε, αναφοράς, κατάθεσης αναφοράς, <clears throat> πρέπει να το έχουν όλοι οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανεξάρτητα από την ηλικία τους. Επαναλαμβάνω, ανεξαρτήτως ηλικίας και δεν έχει γίνει καμία επανάσταση. Εμείς κατορθώσαμε να χειριστούμε ένα σύστημα αναφορών το οποίο είναι ανοιχτό. Νομίζω λοιπόν ότι ε, πάρα πολλοί εδώ στο Κοινοβούλιο αισθάνονται ότι ε, θα πρέπει να κατέβει το όριο, ε, να φτάσει στα 16, αυτό ήδη αναφέρθηκε, μπορούμε να προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο. Γιατί αν πραγματικά επιθυμούμε να επιτρέπουμε τη συμμετοχή, τότε αυτός είναι ο σωστός δρόμος για να γίνει, κυρίως όσον αφορά στους νέους μας. Και στη τελική ανάλυση αυτό που τους λέμε είναι ότι έχετε το δικαίωμα να υπογράφετε. Αυτό ε, μπορεί να είναι ε, πρώτη άσκηση δημοκρατικού σας δικαιώματος, αργότερα μπορείτε και να ψηφίσετε. Επίσης αισθανόμαστε ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με μια ευρωπαϊκή ε, πρωτοβουλία πολιτών. Ε, αν λοιπόν έχουμε διαφορετικές ηλικίε και διαφορετικά δικαιώματα, τότε αυτομάτως ε, θα υπονομεύσουμε την κατάσταση και δεν θα έχουμε ίσους όρους συμμετοχής. Και υπάρχει και ένα άλλο θέμα που θέλω να αναφέρω. Πώς μπορούμε να ελέγχουμε τις υπογραφές. Πράγματι είναι αλήθεια ότι θα πρέπει να συμμετέχουν όλα τα κράτη-μέλη στην επαλήθευση ε, των υπογραφών. Όμως, ε, αν κάποια κράτη-μέλη αρχίσουν να ερωτούν και καταλαβαίνω ότι αυτό μπορεί να συμβεί σε ορισμένα κράτη-μέλη, αρχίσουν να ζητούν ε, ταυτότητες, ε, διαβατήρια. Αυτό μπορεί να είναι ανα, ανατρεπτικός, ανασταλτικός παράγον και έχουν γίνει ήδη κάποιες έρευνες που δείχνουν ότι πράγματι έτσι θα είναι. Γνωρίζουμε αρκετά κράτη-μέλη δεν θα ζητήσουν ταυτότητα. Γι' αυτό λοιπόν ε, έκκλησή μας είναι όταν κατατίθεται αναφορά στο Κοινοβούλιο να μην είναι ε, απαραίτητη και η επίδειξη της ταυτότητας. Γιατί να πρέπει κανείς να δείξει ταυτότητά του αν πρέπει να υπογράψει. Ας προσπαθήσουμε να ε, παραμείνουμε με όσο λιγότερη γραφειοκρατία γίνεται. Και κάτι άλλο που είναι η εμπειρία μας από την Επιτροπή Αναφορών. Ε, όταν προσφέρει κανείς κάτι στους Ευρωπαίους πολιτές θέλουν ένα αποτέλεσμα, μία απάντηση. Πρέπει λοιπόν να είμαστε απόλυτα σαφείς ότι σε τελική ανάλυση αν έχουν συγκεντρωθεί σωστά χίλιες υπογραφές τότε και η Κομισιόν υποχρεούται να απαντήσει όπως ακριβώς ε, απαντάει στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Αυτό πρέπει να είναι απόλυτα σαφές και οι πολίτες να ξέρουν ακριβώς ποια θα είναι η ανταπόκριση. Προσπελασιμότητα, απλούστευση, ευρωπαϊκό πνεύμα, όλα αυτά θα πρέπει να συνοθούν. Πρόεδρος, Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλλά εντωμεταξύ θα ήθελα και να καλωσορίσω την κυρία Ματσόνη, η οποία έφτασε και είναι πρόεδρος της Επιτροπής Αναφορών. Ε, πολύ σωστά κάθεται εδώ, πάνω σε αυτό το τραπέζι, για να ξέρουμε και ποιος είναι. Τώρα λοιπόν μπορεί να λάβει το λόγο ο κύριος Χέφνερ, γιατί μιλάνε οι συγητές. Και μετά θα αρχίσουν οι δικές μας ε, οι παρεμβάσεις. Ίσως θέλετε τώρα να πείτε όμως ένα μικρό χαιρετισμό κυρία Ματσόνη ή μετά, μετά για να κερδίσουμε χρόνο. Και έχουμε κι άλλη μία αντιπρόεδρο, την κυρία Ρούτεν. Μετά βέβαια θα δώσω το λόγο να μπορούν να παρέμβουν και άλλοι αντιπρόεδροι, όπως ο κύριος Σεύκοβιτς. Σε αυτή τη φάση νομίζω ότι μπορούμε να δώσουμε το λόγο στον κύριο Χέφνερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η πρωτοβουλία Ευρωπαίων ε, πολιτών είναι μία από τις μεγάλες υποσχέσεις που έδωσε η Ευρώπη με τη συνθήκη της Λισαβόνας στους πολίτες της για να γίνει ακριβώς η Ευρώπη αυτή περισσότερο Ευρώπη των πολιτών. Είπε και ο κύριος Λαμασούρ ότι εμείς τα ευρωπαϊκά όργανο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είμαστε μακριά από τους πολίτες και οι πολίτες νιώθουν πολύ μακριά από το χώρο που λαμβάνονται οι αποφάσεις. Έτσι λοιπόν με την ε, πρωτοβουλία αυτή μπορούν να κάνουν οι πολίτες προτάσεις, να δίνουν τις ιδέες τους και να ζητούν έτσι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προχωρήσει σε νέες νομοθετικές διατάξεις. Είναι η πρώτη φορά που έχουμε ένα τέτοιο υπερεθνικό μέσο στη διάθεσή μας. Είναι πολύ σημαντικό και πολύ σημαντικό για την Ευρώπη να δείξει στον κόσμο ότι έχουν και αυτοί λόγο στις Βρυξέλλες. Ανοίγουμε έτσι τις πόρτες στις Βρυξέλλες για τους Ευρωπαίους πολίτες. Αυτή πρέπει να είναι η προσέγγισή μας για να δουλέψουμε πάνω στο ζήτημα. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι είναι σημαντικό. Συνήθω έχουμε έναν εισηγητή ή άντε το πολύ να έχουμε δύο εισηγητέ. Ε, λοιπόν, αυτή τη φορά έχουμε τέσσερι εισηγητέ από τέσσερι διαφορετικέ χώρε και τέσσερι διαφορετικέ πολιτικέ ομάδε. Συνεργαζόμαστε στενά με την Επιτροπή και με το Συμβούλιο για να καταλήξουμε σε ένα καλό αποτέλεσμα. Αλλά λέμε ότι θέλουμε να είμαστε ανοιχτοί. Δεν είναι σίγουρο κατά πόσο η πρωτοβουλία αυτή Ευρωπαίων πολιτών θα ενθαρρύνει τον κόσμο να συμμετέχει περισσότερο στις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Μπορεί να οδηγήσει σε απογοητεύσεις αντίθετα. Αν για παράδειγμα μαζέψουν οι πολίτες ένα εκατομμύριο υπογραφές και τελικά στο τέλος μετά από έξι μήνες πάρουν μια επιστολή από την Επιτροπή που να τους λέει ε, μπράβο ευχαριστούμε πάρα πολύ αλλά δεν θα ακολουθήσουμε την πρότασή σας, καταλαβαίνετε ότι αυτό θα οδηγήσει σε απογοητεύσεις. Δεν φτάνει. Γι' αυτό Πρέπει να φροντίσουμε με τη διαδικασία αυτή να δημιουργηθεί διάλογος ανάμεσα στους πολίτες και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Πάνω σε αυτήν την ιδέα δουλεύουμε εμείς οι τέσσερις εισηγητές, ώστε να έχουμε μία πρόταση που να είναι φιλική προς τους πολίτες και όχι πολύ γραφειοκρατική. Το βασικό στοιχείο είναι ο διάλογος. Δεν είναι δημοψήφισμα. Πρόκειται για προτάσεις. Θα δείξω κάποιες πτυχές. Όπως ήδη είπαμε, προτείναμε να διαγράψουμε αυτό το επιπλέον όριο των 300.000 υπογραφών, όταν πρότεινε η Επιτροπή μετά από αυτό να αποφασίζει για το παραδεκτό ή όχι μιας πρωτοβουλίας. Μα δεν είναι δυνατόν να αφήσουμε τον κόσμο να μαζέψουν 300.000 υπογραφές, να έχει γίνει τόση δουλειά πάνω σε αυτές, να έχουν δημιουργηθεί τόσες προσδοκίες και μετά να πούμε «Stop, δεν μπορείτε» ξαναρχίστε γιατί δεν το έχετε κάνει καλά. Όχι. Θέλουμε η επαλήθευση να γίνεται στην αρχή. Φοβόμαστε βέβαια ότι αν γίνει όπως λέει η πρόταση της Επιτροπής από την άλλη, μπορεί οποιοδήποτε να στείλει ένα email και να πει να ορίστε μια πρωτοβουλία Ευρωπαίων πολιτών και έτσι να καταλήξουμε να παίρνουμε εκατοντάδες τέτοιες πρωτοβουλίες που να μην είναι σοβαρές. Πρέπει να βρεθεί λοιπόν ένας τρόπος και είπαμε να είναι 7 πολίτες από 7 διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες. Που σημαίνει ότι θα το έχουν σκεφτεί σοβαρά, ότι θα πρόκειται για σοβαρούς ανθρώπους που έχουν σκεφτεί, έχουν οργανωθεί και μετά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ελέγξει. Είναι αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μήπως είναι κάτι το οποίο αντιβαίνει στις συνθήκες. Και μετά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πει ναι, μπορείτε να αρχίσετε να συγκεντρώνετε υπογραφές. Για την επαλήθευση τώρα των δηλώσεων αυτών υποστήριξη των υπογραφών. Το είπε και η Νταϊάννα, αλλά εγώ θέλω να προσθέσω δύο εδώ. Το ένα είναι το χρονοδιάγραμμα. Εμεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν βλέπουμε γιατί να έχουμε μια μικρή προθεσμία 12 μήνη. Στις χώρες μέλη μπορεί να φτάνει, αλλά σε ευρωπαϊκό επίπεδο αν θέλεις να μαζέψεις υπογραφές από πολλές χώρες μέλη, δεν φτάνει το 12 μήνο και δεν θέλουμε να πιεστούμε, δεν θέλουμε να πιέσουμε τον κόσμο και τελικά μόνο λίγοι ή ορισμένες μεγάλες οργανώσεις στην Ευρώπη να μπορούν να συμμετέχουν. Όχι, εμείς θέλουμε όλες οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις να είναι ενήμερες και να έχουν την ευκαιρία να συγκεντρώσουν υπογραφές. Γι' αυτό εμείς προτιμάμε 18 μήνες προθεσμία και όχι 12. Τέλος, το μεγάλο θέμα. Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στην Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών και τις αναφορές. Ή, για να το πω αλλιώς, για ένα εκατομμύριο υπογραφές. Τι παίρνουν οι πολίτες, αν είναι να πάρουν μια επιστολή μετά, δεν φτάνει. Γι' αυτό προτείνουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι υποχρεωμένη να καλέσει τους πολίτες για μια δημόσια κρόαση, να τους ακούσει, να ακούσει τα επιχείρηματά τους. Πάλι εδώ βρισκόμαστε στην ιδέα που λέει ανοιχτές πόρτες, διάλογος με τους πολίτες. Έτσι θα μπορούσε να αποδώσει τα μέγιστη πρωτοβουλία Ευρωπαίων πολιτών είναι η Ευρώπη μας, πρέπει να καταλάβουν οι πολίτες, μπορούμε να τις κάνουμε, να κάνουμε προτάσεις σε αυτή την Ευρώπη και να υπάρχει κάποια συνέχεια. Αν μη τι άλλο λοιπόν, να είμαστε υποχρεωμένοι να τους ακούσουμε, να τους πάρουμε στα σοβαρά. Ευχαριστώ. Thank you, uh, Mr. And, um, Ευχαριστώ. Κι εγώ ε, συμφωνώ με την λογική αυτή απόλυτα. Από τη Γερμανία τώρα, ε, Ροτ, έχετε το λόγο, παρακαλώ. Ε, Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, πρώτα απ' όλα σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε τη δυνατότητα σήμερα να σας παρουσιάσω την άποψη του Bundestag της Γερμανίας. Ε, βεβαίως και να ακούσουμε και την άποψη των υπολείπων εθνικών κοινοβουλίων. Εγώ αισθάνομαι ότι είναι μεγάλη τιμή αυτό για μένα και ελπίζω να μπορέσω και εγώ να συνεισφέρω στη συζήτηση. Κατά τη δική μας λοιπόν άποψη, η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών θα πρέπει πρώτα απ' όλα να εξυπηρετεί την Ευρώπη. Για μας λοιπόν αυτό σημαίνει ότι χρειαζόμαστε μια ε, φιλική προς τον πολίτη, όχι μη γραφειοκρατική ε, και έγκαιρη πρωτοβουλία, στην οποία θα συμβάλλουν όλοι. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, αλλά και τα Εθνικά Κοινοβούλια καλούνται να βοηθήσουν, γιατί με τις εθνικές τους ε, κυβερνήσεις αυτή τη στιγμή ε, βρίσκονται σε διάλογο οι βουλευτές που βρίσκονται σήμερα εδώ ε, είναι οι εταίροι των πολιτών. Γι' αυτό λοιπόν και δικό μας καθήκον είναι ε, σε αυτή την όλη ε, διαδικασία να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες του πολίτη. Αυτό που μας χαροποιεί ιδιαίτερα και ευχαριστώ για αυτό το λόγο θερμά τους εισηγητές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ευχαριστώ λοιπόν όλους ε, για το ότι τελικά μοιάζει να επικρατεί συνένεση τουλάχιστον ε, κατά την άποψη πολλών συναδέλφων του Κοινοβουλίου της Γερμανίας. Μέχρι τώρα είχαμε δύο συζητήσεις στο Bundestag για την πρωτοβουλία των πολιτών και κατατέθηκε μία σειρά ε, προτάσεων από την αντιπολίτευση και η δική μου η πολιτική ομάδα εκμεταλλεύθηκε τη διαδικασία διαβουλεύσεων για να τοποθετηθεί και αυτή. Βεβαίως δεν θα πρέπει να υπερβάλλουμε ως προς την πολιτεία ε, πρωτοβουλία των πολιτών γιατί αποτελεί συμπλήρωμα της δημοκρατίας. Όμως όλοι μας αισθανόμαστε ότι χρειαζόμαστε περισσότερη δημοκρατία στην Ευρώπη και πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη μας τους πολίτες πρέπει να εξευρωπαίσουμε τους, ε, τις συζητήσεις, ε, τους ε, οργανισμούς, τα κόμματα. Αυτό που διαπιστώνω και με ανησυχεί πάρα πολύ είναι ότι αυτή τη στιγμή βιώνουμε τάσεις επανεθνικοποίησης. Λαϊκίστικα κόμματα που θέλουν να αποκοπούν από την Ευρώπη. Τα κόμματα αυτά κερδίζουν έδαφος συνεχώς Πρέπει όμως να ρίξουμε τα τύχη, τύχη και όχι να ορθώσουμε καινούρια, ε, να δημιουργήσουμε γέφυρες. Έτσι λοιπόν μια πρωτοβουλία η οποία δεν αναλαμβάνεται από κράτος μέλος ή από πολιτικό κόμμα ή από εθνικό οργανισμό αλλά μια πρωτοβουλία που έρχεται από την καρδιά της Ευρώπης αυτή σίγουρα θα βοηθήσει. Ε, δεν πρέπει ούτε να υπερτιμάμε, αλλά ούτε και να υποτιμάμε το εργαλείο αυτό. Εμένα, με ενοχλούν αντιδράσεις ε, που εκφράζονται. Αυτό το είπε και ο συνάδελφος κύριος Χέφνερ και όλοι οι προλαλήσαντες. Δεν πρόκειται για δημοψήφισμα, πρόκειται για πρωτοβουλία. Αλλά ε, μια τέτοια πρωτοβουλία πρέπει να ληφθεί σοβαρά από όλα τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα να αναφέρω και κάποιες άλλες προσδοκίες του Γερμανικού Κοινοβουλίου, ε, γιατί νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό τελικά συμπίπτουν οι απόψεις μας και αυτό εμένα με κάνει ιδιαίτερα αισιόδοξο. Εμείς προσδοκούμε ότι αυτό που παλαιότερα έλεγε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, το 1 τρίτο των κρατών μελών, εμείς λέμε το 1 τέταρτο των κρατών μελών θα πρέπει να αρκεί ως ε, κατώτατο όριο. Επίσης ε, η απαρτία και αυτή ρυθμιστήκε με μεγαλύτερη ευελιξία. Να δούμε στην πράξη, στα κρατημέλη, τέτοιου είδους αναφορές ή πρωτοβουλίες πόσο σοβαρά λαμβάνουν υπόψη από τους πολίτες. Τώρα, ε, ο έλεγχος, μάλλον η έγκρισή μας και η διαδικασία που γίνεται για να δοθεί, αυτή πρέπει να γίνεται στην αρχή. Γιατί είναι παράλογο ε, εκατοντάδε πολιτών να δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο μιας πρωτοβουλία και μετά να τους λέμε ότι ξέρετε αυτό δεν είναι ελπιδοφόρο διότι η, δεν υπάρχει καν αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό οδηγεί σε μεγαλύτερη απογοήτευση και οπωσδήποτε ε, προκαλεί σκεπτικισμό στην Ευρώπη. Ε, γι' αυτό όλα αυτά να εξεταστούν ευθύ εξ αρχής. Εξάλλου, δεν πρέπει να υπάρχουν και άλλοι οργανισμοί ε, για την ε, χορήγηση της ε, άδειας, για την έγκρισή μας. Υπάρχουν, υπάρχει μια σειρά σοφών, αυτοί μπορούν να επιληφθούν του θέματος και εγώ σκέπτομαι γιατί δεν αναθέτουμε στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να συμπεριληφθεί σε αυτή τη διαδικασία. Ε, μπορεί να είναι και άλλη επιτροπή, εγώ δεν θέλω να ανακατευτώ, όμως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να παίζει ρόλο η Κομισιόν αναγκαστικά λόγω της συνθήκης της Λισαβόνας έτσι και αλλιώς παίζει σημαντικό ρόλο, δεν δείτε θέμα επ' αυτού. Δεν χρειαζόμαστε λοιπόν καινούργια όργανα να περιοριστούμε σε αυτά τα οποία ήδη υφίστανται. Επίσης, εμείς ε, θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρχει και το δικαίωμα ε, κατάθεσης έφεσης, διότι οι πολίτες ε, οι οποίοι αναλαμβάνουν μια τέτοια πρωτοβουλία ενδέχεται να μην ε, συμφωνούν με μια απόφαση της Κομισιόν, να μπορούν να καταθέσουν προσφυγή. Ε, το δικαίωμα κατάθεση προσφυγής ε, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Και αυτό που με χαροποιεί ιδιαίτερα είναι η όλη συζήτηση να είναι προσανατολισμένη προς την πρακτική εφαρμογή. Να εκπονηθούν κατευθυντήριες γραμμές για όσους επιθυμούν να αναλάβουν πρωτοβουλίες και αυτό σίγουρα ε, θα συμβάλλει στο να βρούμε μία λύση φιλική προς τον πολίτη. Σήμερα βεβαίως ε, είναι αδύνατο να μην χρησιμοποιεί κανείς τα επιγραμμικά μέσα. Και γι' αυτό ίσως πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη διαδικασία την online, την επιγραμμική, ε, που βέβαια πολλούς πολίτες τους φοβίζει. Το γερμανικό Bundestag εδώ και πολύ καιρό έχει ένα σύστημα κατάθεσης αναφορών online και εγώ θεωρώ ότι είναι απαραίτητο Μάλλον, εγώ θεωρώ ότι τελικά, αν ένα πολίτη αναφέρει το όνομά του και τη διεύθυνσή του, δεν χρειάζεται να αναφέρει και τον αριθμό τη ταυτότητά του. Τουλάχιστον σε εμά το Bundestag, μπορεί κανεί να καταθέσει αναφορά με το όνομα και τη διεύθυνση χωρί αριθμό ταυτότητα. Γιατί λοιπόν εδώ στην Ευρώπη να δημιουργούμε ε, περισσότερε δυσκολίες και απαιτήσει από ό,τι στα εθνικά κοινοβούλια. Εξάλλου, χαιρετίζω το ότι οι εισηγητές προτείνουν διάλογο ε, πριν γίνει ε, ο τελικός, ε, πριν ολοκληρωθεί μια διαδικασία. Αν όλοι αυτοί έχουν, κάνει τόσ, έχουν αναλάβει μεγάλες προσπάθειες, κατέβηκαν στους δρόμους, μάζεψαν πρωτοβουλίες, θα πρέπει, εν πάση περιπτώσει, να έχουν το δικαίωμα να ξεκινήσουν διάλογο με την Κομισιόν. Αναφέρθηκε επίσης και το θέμα του χρονοδιαγράμματος. Εγώ τάσομαι υπέρ ρεαλιστικής λύσης. Κατά την άποψή μου, οι 12 μήνες δεν αρκούν. Οι 18 μήνες σε μια πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία βεβαίως και αρκούν ως χρονικό διάστημα και πριν την εκπνοή αυτού του διαστήματος, αν έχει επιτευχθεί ο στόχος το 1 εκατομμύριο υπογραφές, τότε μπορεί ε, το, ε, η διαδικασία να ολοκληρωθεί χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση. Δηλαδή όταν θα μαζεύονται το 1 εκατομμύριο υπογραφές να κλείνει πιο γρήγορα η διαδικασία. Κατόπιν τούτου, παρακαλώ, τόσο το Συμβούλιο όσο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ολοκληρώσουν το στομότερο δυνατόν τη διαδικασία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δείξει ότι παίρνει σοβαρά υπόψη της τους πολίτες, ότι δεν φοβάται την πρωτοβουλία, κάθε άλλο χαίρεται για αυτήν και επιθυμεί ε, στο μέλλον όλων να αντιμετωπιστούν με σοβαρότητα. Γι' αυτό λοιπόν αγαπητοί συνάδελφοι να προχωρήσουμε στις διαβουλεύσεις μας και να ολοκληρωθούν κατευχήν τα πράγματα. Εγώ αυτό εύχομαι. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πολύ. Ας προσπαθήσουμε να συμπληρώσουμε την πρώτη αυτή φάση, το πρώτο αυτό τμήμα της συζήτησης. Ακούγοντας πλέον μετά από τους τέσσερις συζητητές και μετά από την κυρία Ρίτεν, η οποία παρουσίασε συμφετικά τις απόψεις των κοινοβουλίων των κρατών μελών τον κύριο Ολιβιέ Σαστέλ, Προεδρεύοντα του Συμβουλίου. Κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, και οι συνάδελφοι από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Κοινοβούλια των Κρατών Μελών να πω όπως και πάρα πολλοί άλλοι ότι ένα από τα βασικά βήματα προς τα εμπρός της συνθήκης της Λισαβόνας είναι η ενίσχυση του δημοκρατικού χαρακτήρα της Δημοκρατικής Ένωσης με διαφορετικές μορφές ενίσχυση των αρμοδιοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, περαιτέρω εμπλοκή των κοινοβουλίων των κρατών μελών στην Ευρωπαϊκή Διαδικασία Λήψης Αποφάσεων, σημαντική ενίσχυση της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας και όπως άλλοι είπαν πριν από μένα, ξεκινώντας με τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου, η συνθήκη της Λισαβόνας, του Βελγίου εννοώ, διευρύνει τη συνεργασία με τους πολίτες, συνδέει τον πολίτη μέσω της δημοκρατίας της αντιπροσωπευτικής με επιπλέον μέσα και εδώ έρχεται το δικαίωμα πρωτοβουλίας των πολιτών που θα επιτρέψει στον πολίτη να οδηγεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει προτάσεις νομοθετικές. Πρόκειται για από τις πιο θα έλεγα συγκεκριμένες πλευρές των καινοτοπιών της συνθήκης της Λισαβόνας. Κάτι τέτοιο θα διευκολύνει την συζήτηση τη διασυνοριακή και την εμφάνιση ενός πραγματικού ευρωπαϊκού χώρου. Γι' αυτό ακριβώς χαίρομαι που είμαι ανάμεσά σας σήμερα για να ακούσω τις απόψεις σας. Είμαι σίγουρος ότι οι απόψεις σας είναι τμήμα των ανταλλαγών θέσεων που έχουμε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στα πλαίσια της εφαρμογής αυτού του δικαιώματος απαιτείται να βρεθεί μια ισορροπία. Μια ισορροπία όχι εύκολη. Οι κανόνες και οι διαδικασίες δεν μπορεί να είναι αποκλειστικά αποτρεπτικές. Το μέσο θα πρέπει να είναι κοντά στον Ευρωπαίο πολίτη και θα πρέπει να είναι εύκολο στον τρόπο με τον οποίο θα το πλησιάσει ο πολίτης. Θα πρέπει να δει διεγγυήσεις και για την αξιοπιστία του ονομοθέτης. Το Συμβούλιο, όπως γνωρίζετε, ήδη από την 14η Ιουνίου, εδώ και τρεις περίπου μήνες, κατέληξε σε ορισμένες γενικές κατευθύνσεις για την πρόταση ε, ε, κανονισμού σχετικά με την εφαρμογή της νέας αυτής μεθόδου. Δεν θα μπω σε τεχνικές λεπτομέρειες, θα σας θυμίσω όμως κάποια στοιχεία αυτού του προσανατολιστικού κειμένου. Το Συμβούλιο προτείνει να ορίσει τον ελάχιστο αριθμό κρατών από όπου πρέπει να προέρχονται οι υπογραφές στο 1 τρίτο των κρατών μελών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά να υπάρξει επίσης και ένας ελάχιστος αριθμός πολιτών ανά κράτο μέλος επί τη βάση ενός μαθηματικού τύπου που θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των ευρωβουλευτών κάθε χώρας και έτσι ο κατώτερος αριθμός δεν ήταν το, το επίπεδο ελέγχου και αποδεκτού ημί της πρωτοβουλίας δεν είναι 300.000 αλλά 100.000. Οι πρωτοβουλίες οι οποίες δεν εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής της συνθήκης βέβαια είναι υβριστικές, δεν είναι σοβαρές ή είναι ενάντιες στις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να απορρίπτονται άμα τη καταγραφή τους. Ο κανονισμός, η πρόταση κανονισμού μάλλον ζητάει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προχωρήσει στην δημιουργία ενός λογισμικού το οποίο να είναι ελευθέρας πρόσβασης για την συλλογή υπογραφών online. Ένα τέτοιο λογισμικό θα επιτρέψει στους οργανωτές των πρωτοβουλειών αυτό να ξεκινήσουν τις πρωτοβουλίες τους πιο εύκολα, σεβόμενοι πάντα τους βασικούς κανόνες προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Τέλος, το Συμβούλιο διευκρινίζει την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής λέγοντας ότι για κάθε κράτος μέλος απαιτούνται ε, τα στοιχεία αυτών οι οποίοι υπογράφουν και θα πρέπει δειγματοληπτικά να επαληθεύονται οι υπογραφές αυτές. Αυτό θα επιτρέψει να απαντήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Πού βρισκόμαστε σήμερα λοιπόν δεν θα μιλήσω εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά και στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο, περιμένουμε την τελική θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τις διαπραγματεύσεις σε επίπεδο τριμερούς διαλόγου και να μπορέσουμε να προχωρήσουμε επί τη βάση μιας ημερήσιας διάταξης η οποία να είναι καθορισμένη πλέον και η οποία θεωρητικά θα πρέπει να μας οδηγήσει μέχρι το τέλος του χρόνου στο να έχουμε ορίσει πλέον τους κανονισμούς λειτουργίας αυτού, τους τρόπους λειτουργίας μάλλον αυτού του κανονισμού. Είναι επίγον το θέμα γιατί ήδη την 1η Δεκεμβρίου θα είναι σε ισχύ ε, η συνθήκη της Λισαβόνας για ένα χρόνο και ο πολίτης δεν θα καταλαβαίνει γιατί ένα χρόνο μετά τα τρία όργανα μας συζητούν, τσακώνονται μεταξύ τους για να μπορέσουν ε, να αποφασίσουν και να προτείνουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια σειρά θεμάτων προσυζήτηση. Λοιπόν, εδώ βρισκόμαστε σήμερα. Συνεργαζόμαστε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, έχουμε συναντήσεις συχνές, επικοδομητικές. Ελπίζω ότι θα πρέπει όμως κάποια στιγμή να καταλήξουμε για να μπορέσουμε να επισημοποιήσουμε τους κανόνες οι οποίοι θα ισχύσουν για τη σωστή λειτουργία της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας των πολιτών. Νομίζω ότι είναι ένα από τα πιο δημοκρατικά μέσα τα οποία θέτει στη διάθεση του πολίτη η συνθήκη της Λισαβόνας. Σε ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε για την παρουσίασή σας. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την συνεχή, σταθερή, φιλική επακριβέστατη παρουσία σας στα όργανα αυτού εδώ του Κοινοβουλίου. Λοιπόν, το ίδιο θα πρέπει να πω επίσης και για τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον Μάρο Σεύκοβιτς. Έχει έρθει επανειλημμένα στην Επιτροπή μας ο κύριος Σεύκοβιτς, τον έχουμε ακούσει επανειλημμένα και στην Ολομέλεια και είναι κάποιος ο οποίος ακούει προσεκτικά τις απόψεις του Κοινοβουλίου. Πρόεδρε Σεύκοβιτς, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Εθνικών Κοινοβουλίων. Είναι μεγάλη χαρά για μένα που έχω την ευκαιρία να έρθω εδώ και να συζητήσω μαζί με εσάς και τους Ευρωβουλευτές και τους βουλευτές από τα Εθνικά Κοινοβούλια ένα τόσο σημαντικό θέμα όπως είναι η Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών. Γιατί αν δείτε ποιος κερδίζει από τη συνθήκη της Λισαβόνας, είναι ξεκάθαρο ότι είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα Εθνικά Κοινοβούλια και οι πολίτες οι κερδισμένοι από τη συνθήκη αυτή. Προσπαθούμε όσο περνά ο καιρό να εφαρμόζουμε όλο και περισσότερο και να θέτουμε σε εφαρμογή τι διατάξει τη συνθήκη τη Λισαβόνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ιδιαίτερα τα Εθνικά Κοινοβούλια εκείνα τα οποία συνεισέφεραν τόσο πολύ στην προετοιμασία τη πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών. Βοήθησαν τα σχόλιά σα στην πράσινη βίβλο που ήρθε από την Τσεχία, την Πορτογαλία και την Ιρλανδία όταν ε, ετοιμάζαμε το σχέδιό μας για να ε, οδηγηθούμε στην πρωτοβουλία Ευρωπαίων ε, πολιτών. Και η Κύπρος επίσης, όταν το σχέδιο είχε ετοιμαστεί, βοήθησαν για να μας κατευθύνουν στις μελλοντικέ μας συζητήσεις με το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είμαστε υπόχρεστο στο Συμβούλιο για την εξαίρετη συνεργασία που είχαμε μαζί του, όπως επίσης και στην Ισπανική Προεδρία που ήταν πολύ επικοδομητική. Και η Βέλγικη είναι εξίσου επικοδομητική τώρα. Έτσι μπορούμε, πιστεύω, πολύ σύντομα να καταλήξουμε σε μια συμφωνία, λίγους μήνες δηλαδή, μετά την αρχική πρόταση της Επιτροπής για την Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών. Εννοείται ότι τώρα περιμένουμε την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από ό,τι άκουσα θα είναι έτοιμη πολύ σύντομα. Τότε θα μπορέσουμε να προωθήσουμε ακόμα περισσότερο την πρόταση αυτή και να τη συζητήσουμε στον τριμερή διάλογο. Περισσότερες από τις λεπτομέρειες τις ακούσαμε από τον κύριο Σαστέλ. Άκουσα επίσης τον κύριο Ρώτα από την Bundestag πολύ προσεκτικά και διαπιστώνω ότι υπάρχει σύμπτωση απόψεων ανάμεσα στην Πούτεστακ και στους συναδέρφους από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επιτρέψτε μου τώρα να σας εξηγήσω λιγάκι πώς βλέπουμε εμείς αυτά τα θέματα τα οποία τόσο ωραία παρουσίασαν οι προηγούμενοι ομιλητές. Ένα τρίτο των κρατών μελών. Αυτό είναι το πρώτο θέμα. Γιατί αποφασίσαμε το ένα τρίτο. Γιατί θεωρήσαμε ότι ήταν λογικό να έχουμε το 1 τρίτο των χωρών μελών και να έρχονται οι υπογραφές από το 1 τρίτο των χωρών. Γιατί, γιατί αυτό το 1 τρίτο πιστεύουμε ότι είναι ένα στοιχείο κλειδί για να έχουμε και την ενισχυμένη συνεργασία και για να ξεκινήσει η επικουρικότητα, ο έλεγχος της επικουρικότητας. Κάθε φορά μιλάμε για το 1 τρίτο των χωρών. Επίσης, θέλαμε η πρωτοβουλία Ευρωπαίων πολιτών να είναι πραγματικά ευρωπαϊκή, δηλαδή να έχει ευρωπαϊκό χαρακτήρα. Και πώς θα το ξέρουμε αυτό, αν δεν έχουμε πρωτοβουλίες τοπικού ή περιφερειακού χαρακτήρα, γι' αυτό θελήσαμε το 1 τρίτο Έχουμε υπόψη μας ότι οι πρωτοβουλίες που έρχονται από ένα τρίτο των χωρών μελών θα ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προχωρήσει σε νομοθετική πρόταση που θα πρέπει να εφαρμοστεί και στις 27 χώρες μέλη. Γι' αυτό πρέπει να έχει ευρωπαϊκή διάσταση η πρωτοβουλία ευθύ εξ αρχής. Και χαίρομαι που ο κύριος Ροτ συμφωνεί με την αλλαγή που κάναμε στον υπολογισμό πώς υπολογίσουμε δηλαδή τον αριθμό των υπογραφών που χρειαζόμαστε από κάθε κράτος μέλος. Ακούσαμε πράγματι τις ε, γερμανικές ανησυχίες που εισακούστηκαν ουσιαστικά και έτσι μιλάμε για το 0,2% του πληθυσμού για τη Γερμανία. Θα χρειάζεται 160.000 υπογραφές. Και μόνο χίλιες υπογραφές χρειαζόμαστε από το Λουξεμβούργο με το νέο αυτό υπολογισμό όπου λάβαμε υπόψη μας τον ε, αριθμό των χωρών και πόσους κατοίκους έχει κάθε χώρα. Έτσι δεν αποκλείονται ούτε οι μεγάλες χώρες, αλλά και αυτές μπορούν πιο εύκολα να συμμετέχουν στην δημοκρατική αυτή διαδικασία. Ένα άλλο θέμα που πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους νέους είναι το εξή. Αποφασίσαμε και είναι το πρώτο δημοκρατικό μέσο αυτό στην Ευρώπη, ίσως εκτός από την Εστονία, που επιτρέπουμε online συλλογή υπογραφών, συγκέντρωση υπογραφών. Είναι βέβαια μια σύγχρονη προσέγγιση. Είναι έτσι πιο εύκολη η συγκέντρωση των ε, υπογραφών, πιο εύκολη, κινητοποιούνται περισσότερο οι πολίτες αλλά βέβαια υπάρχει και κάποιος κίνδυνος συγχρόνως, ε, που είναι η προστασία των προσωπικών δεδομένων και ο ελεγχός τους. Αλλά παρόλα αυτά θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τη σύγχρονη τεχνολογία για να μπορέσει έτσι να κινητοποιηθεί πιο εύκολα ο κόσμος. Επίσης κοιτάξαμε πάρα πολύ καλά τις συστάσεις του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το software, το πρόγραμμα. Να δούμε δηλαδή πώς μπορούμε να έχουμε ένα πρόγραμμα ανοιχτής πηγής, open source, ώστε να μην χρειάζεται η πιστοποίηση που θα έπρεπε να φροντίσουν γι' αυτό οι ίδιοι οργανωτές και θα ήταν μια πολύ πιο βαριά διαδικασία. Τώρα θα υπάρχει μια ανοιχτή πηγή και έτσι θα είναι πιο εύκολα τα πράγματα για τους διοργανωτές. Τώρα το στο θέμα του παραδεκτού της ε, πρωτοβουλίας. Από τη μια, θέλουμε να ενθαρρύνουμε τους πολίτες να συμμετέχουν στη δημοκρατική ζωή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εντάξει. Από την άλλη μεριά, έχουμε αρκετή εμπειρία με καταχρήσεις τέτοιων συστημάτων. Γίνεται αρνητική προπαγάνδα, υπάρχουν πρωτοβουλίε που αντιτίθεται στι αξίε και τι αρχέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αντιτίθεται στα ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι πρωτοβουλίε επιπόλε, έτσι ελαφρέ και όχι Γι' αυτό θέλουμε μια πλατφόρμα που να χρησιμοποιείται για το σκοπό για τον οποίο έχουν φτιαχτεί. Και όχι για την αυτοπροβολή κάποιων που θέλουν να ξεκινήσουν μια δύσκολη πολιτική συζήτηση χωρίς καμία πολιτική στήριξη από πίσω. Αλλά και εδώ έχουμε τον άτυπο τριμερή διάλογο με τους Ευρωβουλευτές και τον Υπουργό Σαστέλ και πιστεύω ότι πηγαίνουμε προς μία κατεύθυνση όπου θα βρούμε την καταλληλότερη λύση. Σας διαβαίνω από τη δικιά μας την πλευρά θα φροντίσουμε για την σωστή λύση. Απλώς δεν θέλουμε ένα σύστημα το οποίο θα ξεκινάει όλο το μηχανισμό στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα χρειάζεται και οι επίτροποι να αποφασίσουν. Είναι πολύ δύσκολο να έχουμε ένα τέτοιο σύστημα και γι' αυτό σκεφτόμαστε να αλλάξει λιγάκι η διαδικασία καταχώρησης της πρωτοβουλίας και να βασίζεται σε διοικητική απόφαση. Δεν θα δεχόμαστε πρωτοβουλίες που είναι επιπόλες και όχι που είναι κατά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που δεν επίπτωσαν αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τέτοιες δεν καταχωρούνται. Χτες στην Επιτροπή Αναφορών άκουσα ερωτήσεις που λέγανε καλά και πώς θα ότι αυτό θα γίνεται σωστά. Μα πάντα υπάρχει δυνατότητα οι πολίτες να μπορούν να προσφύγουν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Αν κάποιος πιστεύει ότι εμείς κακώς αποφασίσαμε αυτό που αποφασίσαμε, μπορεί να διορθωθεί η απόφασή μας. Υπάρχει πάντα η δυνατότητα της προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και επιπλέον θα προσφέρουμε στους διοργανωτές ένα help desk που θα μπορούν δηλαδή οι διοργανωτέ να έρχονται σε εμά και να τους δίνουμε βοήθεια, κατευθυντήριες γραμμές για το πώς να βάλουν μπρο την διαδικασία για την υποβολή πρωτοβουλία και κατά πόσο η πρωτοβουλία αυτή εμπίπτει όντως στις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επιτρέψτε μου τώρα, Πρόεδρε, μια τελευταία παρατήρηση. Ας πούμε ότι έχουμε το 1 εκατομμύριο υπογραφές. Τα κράτη-μέλη πρέπει να τις ελέγξουν. Σε τέσσερις μήνες μετά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εκδίδει μία ανακοίνωση για κάθε πρωτοβουλία. Να σας πω ποιες θα είναι οι προθέσεις μας. Τι θέλουμε να κάνουμε και τι διαδικασία θα ακολουθήσουμε. Θα ενημερώνουμε και το Κοινοβούλιο και τις οργανωτές και το Συμβούλιο για κάθε περίπτωση και φυσικά και πρέπει να βελτιωθεί η σύνδεση με τον πολίτη και η ποιότητα της πολιτικής συζήτησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό, γι' αυτό η ιδέα για μια ακρόαση με τους διοργανωτές της εκάστοτε Πρωτοβουλία είναι κάτι θετικό. Δεν ξέρω τώρα αν θα το οργανώνει αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή η Κομισιόν. Σημαντικό είναι να γίνεται συζήτηση με τους διοργανωτές οι οποίοι να έρχονται και να παρουσιάζουν την επιχειρηματολογία τους πως βλέπουν την ε, διαδικασία συλλογής υπογραφών και την όλη συνέχεια. Τέλος, ελπίζω ότι το μέσο αυτό και χαίρομαι που είναι εδώ και τα Εθνικά Κοινοβούλια. Πιστεύω λοιπόν ότι έτσι θα μπορέσουμε να διευρύνουμε την πολιτική συζήτηση στην Ευρώπη και να την φέρουμε πιο κοντά στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Έτσι θα συζητηθεί περισσότερο η Ευρώπη στις εθνικές πρωτεύουσε. Και ελπίζω ότι την επόμενη φορά που θα υπάρξουν ευρωεκλογέ δεν θα κυριαρχούν τα εθνικά ζητήματα σε αυτές, αλλά θα υπάρχουν και περισσότερα ευρωπαϊκά συζήματα που θα απασχολήσουν τότε τους πολίτες μας. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τις σχέσεις των πολιτών με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς ε, και τώρα λοιπόν περνάμε στη δεύτερη φάση ε, στην οποία ε, θα προεδρεύσει η συμπρόεδρος κυρία Ρούτεν. Έχουμε λοιπόν τον κατάλογο των ομιλητών και πρώτα απ' όλα θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Κρούμοβα η οποία εκπροσωπεί την Εθνική Συνέλευση της Βουλγαρίας. Έχετε το λόγο. Πρώτα απ' όλα θέλω να σας πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ που μου δίνετε το λόγο ως πρώτη παρεμβαίνουσα Εμείς θεωρούμε ότι η πρωτοβουλία των πολιτών είναι πολύ σημαντικό εργαλείο για την ενίσχυση της δημοκρατίας, για την μείωση του δημοκρατικού ελλείμματος. Θεωρούμε λοιπόν ότι με αυτόν τον τρόπο οι πολίτες της Ευρώπης μπορούν να ταυτιστούν καλύτερα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσον αφορά τώρα στο οικονομικό βάρος για τα κράτη-μέλη, ε, το βάρος αυτό μπορεί να περιστεί στο ελάχιστο, βεβαίως λαμβάνοντας υπόψη τα δικαιώματα όλων των πολιτών. οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, θα συμμετάσχουν με μεγάλη τους ε, χαρά στην πρωτοβουλία πολιτών εφόσον πρόκειται για κάτι που αφορά παραδείγματος χάρη στη ζωή τους. Είναι πολύ σημαντικό ε, το ότι αποφασίστηκε το 1 τρίτο των κρατών μελών. Αυτός είναι και ο σωστός αριθμός κατά τη γνώμη μου. Και είναι και μια σωστή προσέγγιση. Στη δική μας λοιπόν τη γνωμοδότηση αναφερόμεθα ε, με θετικά σχόλια ε, για το online μητρό στο οποίο θα περιλαμβάνονται όλες οι πρωτοβουλίες των πολιτών και πιο συγκεκριμένα σε όλες τις ευρωπαϊκές γλώσσες. Τελειώνοντας, θα ήθελα να επισημάνω ότι τα αποτελέσματα αυτής της ε, διακοινοβουλευτικής ε, συνάντησης ε, θα συμβάλλουν στην βελτίωση της διαδικασίας, στην ώστε δυνατόν ταχύτερη εφαρμογή αυτού του κανονισμού. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Και εμείς ευχαριστούμε. Πάμε από τη Βουλγαρία ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο, ε, στη Βουλή των Λόρδων, Λόρδος Πόμς. Ευχαριστώ πάρα πολύ και σας και τους συναδέλφους στις... Ε, Πρέπει να πω ότι η υποπιτροπή μας κοίταξε την πράσινη βίβλο και κατέληξε στο συμπέρασμα το ίδιο, το οποίο λίγο πολύ είπαν και άλλοι ομιλητέ σήμερα το απόγευμα, ότι πρέπει να υπάρχει ευρία πρόσβαση του κοινού στη διαδικασία, ότι πρέπει να χρησιμοποιούμε πλήρω το διαδίκτυο, ότι πρέπει να υπάρχει ίση μεταχείριση των χωρών μελών, να υπάρχει όσο γίνεται πιο λίγη γραφειοκρατία, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για, την, για τον έλεγχο των ε, υπογραφών που έχουν συγκεντρωθεί. Σίγουρα χρειάζονται κάποια μέτρα ώστε δεν πρέπει να κάνουν τέτοιες πρωτοβουλίες ομάδες πίεσης. Πρέπει να φροντίσουμε λοιπόν να πετύχουμε όλους αυτούς τους στόχους που έχουν τεθεί. Καταλαβαίνω ότι δεν έχουμε πολύ χρόνο, αλλά να ξέρετε ότι η δικιά μου επιτροπή θα εγκρίνει περίπου 100% τόσο είπε εκπρόσωπος της Bundestag ο κύριος Ροτ. Δεν υπάρχει λόγος να έχουμε τέτοια πρωτοβουλία αν είναι να γίνει τόσο περίπλοκη που τελικά θα φτύει μέσα στη γραφειοκρατία. Ούτε πρέπει να ζητάμε από τους διοργανωτές να φτιάχνουν εκείνοι ιστοσελίδες, ούτε να έχουμε τόσο περίπλοκες διαδικασίες επαλήθευσης. Πρέπει να έχουμε ένα σύστημα που δεν δημιουργεί παρετέρω προβλήματα με προστασία δεδομένων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίσης πρέπει να αποφασίζει πολύ γρήγορα για το παραδεκτό μιας τέτοιας πρωτοβουλίας. Το ένα θέμα που θέλω εγώ να ζητήσω σε σχέση με το έγγραφο εργασίας που έχουμε είναι μία μνήα στην παράγραφο 24.4 στη σελίδα 5 του αγγλικού κειμένου μία πρόταση στο κεφάλαιο που λέει εάν αποφασίσει να μην κάνει νομοθετική πρόθεση, πρόταση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εγώ θα έλεγα να μπορεί να γίνει προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Έτσι λέει μάλλον εδώ. Καταλαβαίνω γιατί το λέτε αυτό. Θα αποφασίσει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, για παράδειγμα, ότι οι διαδικασίες δεν έχουν ακολουθηθεί σωστά, ότι έχει ληφθεί στραβή απόφαση και θα αποφασίσει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ότι κάτι πρέπει παρόλα αυτά να καταχωρηθεί. Όμω, επειδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή της αλλιώ έχει το δικαίωμα πρωτοβουλία, δεν θα πρέπει να υποβάλλεται στη δικαιοδοσία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πρέπει να παραμείνει μια απλή διαδικασία, γιατί αλλιώς θα γίνει πολύ περίπλοκη αν εμπλέκεται και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ναι, να μπορεί να αποφανθεί επί της διαδικασίας, εφόσον γίνουν διαδικαστικά λάθη, αλλά επί της ουσίας δεν πιστεύω ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θα πρέπει να αποφασίσει να ερευνήσει κατά πόσο σωστά ή όχι αποφάσισε να δώσει συνέχεια ή όχι σε μια τέτοια πρωτοβουλία επιτροπή. Υπάρχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια που θα φροντίσουν και τα κράτη-μέλη θα φροντίσουν να δώσει το Συμβούλιο κάποια συνέχεια. Πολύ ωραία, λέει ο Πρόεδρος. Ε, νομίζω ότι αυτή η τελευταία παρατήρηση είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και πιστεύω ότι η Επιτροπή, ασκώντας ε, το δικαίωμά της ε, πρωτοβουλίας, θα διατηρήσει το δικαίωμα της ε, αξιολόγησης, άρα δηλαδή πρέπει να κάνουμε διαφοροποίηση ανάμεσα στις ε, ε, πρακτικές τακτικές, στις τακτικές και στην άσκηση του πολιτικού δικαιώματος. Στην δεύτερη λοιπόν περίπτωση, στην περίπτωση κατά την οποία η απόφαση είναι μόνο πολιτική, και δεν μπορεί κανείς ε, να προβλέψει το κατά πόσο είναι απαραίτητο να υπάρχει ποιοτική παρέμβαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτό το αναφέρω ως μια ιδέα για το μέλλον. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο ε, στον επόμενο μιλητή, στον κύριο Γκρουνή, ε, συνάδελφος Γκρουνί από την Επιτροπή Αναφορών. Κυρία Γκρουνί. Ναι. Ευχαριστώ θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας σε αυτό το εξαιρετικό μέσο, την πρωτοβουλία των πολιτών. Για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες, γιατί θα μπορέσουν να επηρεάσουν καλύτερα τις αποφάσεις στην Ευρώπη. Βέβαια θα μπορέσουν να δημιουργηθεί και δυσθυμία στην περίπτωση που δεν γίνει αποδεκτή μια τέτοια πρωτοβουλία και εδώ έρχομαι στην εμπειρία μου στην Επιτροπή Αναφορών. Η διαδικασία θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτική σχετικά με την αποδοχή ή όχι μιας τέτοιας πρωτοβουλίας και ιδιαίτερα σχετικά με τον χρόνο ο οποίος θα περάσει από τη στιγμή που θα φτάσει η πρωτοβουλία αυτή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη στιγμή κατά την οποία θα κριθεί αποδεκτή η μη. Γι' αυτό ήμουν και σαφέστατα υπέρ της πρότασης ελέγχου του αποδεκτού από τις 5.000 ε, υπογραφές. Δεν χρειάζεται να περιμένουμε εκατοντάδες χιλιάδες. Δεν θα πρέπει να δίνουμε ελπίδες φρούδες στους συμπολίτε μας. Βλέπω σε εξαναφορών ότι λαμβάνουμε πάρα πολλούς αναφορείς οι οποίοι ε, προσδοκούν πολλά και όταν τους απαντούμε αρνητικά, αν ο χρόνος που έχει διαμεσολαβήσει μέχρι την απάντησή μας είναι μεγάλος, τόσο μεγαλύτερη είναι και η απογοήτευσή τους. Συνεπώς λοιπόν δεν θα πρέπει να καλλιεργούμε φρούδες ελπίδες στους πολίτες μας. Δεύτερο, αν δεν θεωρηθεί αποδεκτή μια πρωτοβουλία, αυτό σημαίνει ότι η αναπομπή στην Επιτροπή Αναφορών θα μπορούσε να είναι μία από τις πιθανές λύσεις, εναλλακτικέ λύσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Γκρινή. Ο κύριος Γκλογκόσκι έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Χαίρομαι που τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, η Επιτροπή, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν ξεκινήσει να εργάζονται στα πλαίσια αυτής της πρωτοβουλίας. Στα πλαίσια της επικύρωσης της διαδικασίας της Συνθήκης της Λισαβόνας, το θέμα αυτό συζητήθηκε επί μακρόν και χαρακτηρίστηκε σαν μία από τις βασικές νέες αξίες, θα έλεγα, με ευρωπαϊκή διάσταση. Είμαι βέβαιος ότι όλα αυτά θα συνεισφέρουν στη συζήτηση την οποία είχαμε και νωρίτερα. Να υπάρξει δηλαδή υψηλός βαθμός εμπιστοσύνης των πολιτών μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους θεσμούς της. Είχαμε διαβουλεύσει στην Πολωνία και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υποστηρίξαμε τις περισσότερες από τις προϋποθέσεις που κρίνονται απαραίτητες έτσι ώστε να ξεκινήσει μια τέτοια πρωτοβουλία. E, Εδώ τίθεται και το, θέμα της ηλικία αυτών που μπορούν να παίρνουν μέρος στην διαδικασία. Αυτό είναι κάτι όμως το οποίο μπορεί να αλλάξει έτσι όπως θα συνεχιστούν οι διαδικασίες θα το δούμε ξανά. Ιδιαίτερα θα δούμε τι μπορούν να κάνουν οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι είναι νεότερον, νεότεροι των 18. Τώρα για τους 100.000, για τις υπογραφές όταν φτάσουν τον αριθμό των 100.000. Αυτό στη δική μου χώρα ισχύει μεν, αλλά είναι ένα νέο μέσο και δεν έχουμε συγκεντρώσει πάρα πολλέ εμπειρίες σχετικά με τη λειτουργία του. Πρόκειται για μια καινοτομία δηλαδή και για την χώρα μου γίνονται κάποιες προσπαρασκευαστικές εργασίες σε σχέση με μια νομοθετική ρύθμιση μετά από πρωτοβουλία των Πολωνών πολιτών. Okay, dank u wel. Um, ik heb, uh... Ευχαριστώ 100.000 Ευχαριστώ. Είπατε για 100.000, εδώ μιλάμε για 300.000, υπάρχει βέβαια κάποια διαφορά. Τώρα το λόγο θα έχει ο κύριος Δεμπιάνκη από την Πορτογαλία. Παρακαλώ, από το Πορτογαλικό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Το θέμα της πρωτοβουλίας Ευρωπαίων πολιτών είναι ένα θέμα στο οποίο επιφυλάχτηκε μεγάλο ενδιαφέρον και πολύ θετική αντιμετώπιση στην Πορτογαλία. Είχαμε την δυνατότητα να συζητήσουμε και με τον Αντιπρόεδρο Σέσκοβιτς, ο οποίος μας παρουσίασε την άποψή του σε ένα σεμινάριο που οργανώσαμε στην Εθνική Συνέλευση της Πορτογαλίας. Στη συνέχεια η πρόταση αυτή πήγε στην Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων και στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εννοείται ότι υπάρχουν ε, κάποιες διαφορές. Είναι λογικό μέσα σε ένα κοινοβούλιο όπου εκπροσωπούνται έξι διαφορετικά κόμματα. Παρ' όλα αυτά, διαπιστώσαμε ότι υπάρχει μια πλήρη συνένεση για τα βασικά ζητήματα που περιλαμβάνει η πρόταση αυτή. Το Πορτογαλικό Κοινοβούλιο στην Επιτροπή Σταγματικών Υποθέσεων και στην Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών μάλλον θεμάτων, Ευρωπαϊκών θεμάτων, αποφάνθηκε ξεκάθαρα υπέρ της πρότασης του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Παρ' όλα αυτά, όμως, πιστεύω ότι πρέπει να διαπιστώσουμε ότι κατά τη διάρκεια των συζητήσεων βγήκαν πολλά ζητήματα. Σημειώσαμε μάλιστα την επιφύλαξη όσον αφορά τα κριτήρια του παραδεκτού. Αναφέρθηκε σε αυτό και ο κύριος Λαμασούρ. 100.000, 300.000 και υπάρχουν και κίνδυνοι που ελοχεύουν εδώ και που έχουν να κάνουν με το ότι αν έχουμε ήδη έναν πολύ μεγάλο αριθμό υπογραφών, εφόσον η πρωτοβουλία τελικά δεν κρυθεί παραδεκτή, καταλαβαίνετε τι αίσθηση θα δημιουργήσει στον κόσμο. Όσον αφορά λοιπόν τα διάφορα σημεία στο οποίο αναφέρθηκε ο κύριος Σέσκοβιτς, για την προσφυγή πιο συγκεκριμένα που είπε ο κύριος Σέσκοβιτς, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη μας διάφορες επιφυλάξεις που διατυπώθηκαν εδώ για τους κινδύνους που ελοχεύει κάτι τέτοιο για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κυρίως όσον αφορά τα κριτήρια ε, παραδεκτού ή όχι. Τελειώνω με το εξή. Είναι πολύ σημαντικό η πρωτοβουλία αυτή Ευρωπαίων πολιτών Ακριβώς επειδή οι προϋποθέσεις εκπροσώπησης είναι σημαντικές, αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την ευρωπαϊκή ταυτότητα. Είναι μια πρωτοβουλία η οποία δεν μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο από γραφειοκρατικές υπερβολές κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Προσοχή σε αυτό. Ούτε θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο επικρίσεων όσον αφορά το ευαίσθητο ζήτημα του κατά πόση πρωτοβουλία αυτή μπορεί να κρυθεί παραδεκτή όχι. Ο κύριος Μπρόνς έχει το λόγο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η πρωτοβουλία αυτή ελέγχεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξ Θα πρέπει να συμφωνήσει η Επιτροπή να την κάνει αποδεκτή, να πει αν είναι, ε, θα έλεγα, συμβατή με τις δημοκρατικές αξίες. Τα ίδια γινόντουσαν και στη Σοβιετική Ένωση βέβαια και μετά θα πρέπει για να ελεγχθεί να έχουν ήδη υπογράψει 300.000 και θα ζητηθεί φυσικά η άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ακόμα και όταν φτάσουν οι υπογραφές στο 1 εκατομμύριο. Ε, μπορεί να αρνηθεί πάλι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει οτιδήποτε, δεν προκαλείται αυτόματα δημοψήφισμα, οπότε ο τίτλος «Πρωτοβουλία των πολιτών» δεν είναι σωστός. Νομίζω ότι ένας απλός πολίτης, αν δεν υποστηρίζεται από μεγάλους οργανισμούς, είναι πολύ δύσκολο να φτάσει στο ένα εκατομμύριο από εννέα διαφορετικές χώρες. Είναι κάτι το φανταστικό και μάλιστα κοινικά φανταστικό. Δεν θα υπάρξει επιτυχής πρωτοβουλία και ίσως να περάσουν κάποιες τις οποίες θα προωθούν οι μεγάλες επιχειρήσεις και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η καθεστική ατάξη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ουσία βολεύεται και κάνει τις προτάσεις ε, οι οποίες ακριβώς ε, είναι αυτές που την έχουν εκεί που είναι. Στην περίπτωση που αυτά τα οποία λέγω λάβει κάποιο σοβαρά, τότε ας προκαλέσουν ε, το ένα εκατομμύριο υπογραφές αυτές ένα δημοψήφισμα, ας απομακρυνθούμε από τις σοβιατικές ευρωπαϊκές αξίες, και το θέμα είναι ποιο θα κρίνει ποιε είναι αυτέ οι αξίε. Το να αποφασίζει κανεί ποιε είναι οι αξίε αυτέ, μόνο δημοκρατία δεν είναι. Ehm, eh, Ευχαριστούμε. Το λόγο έχει τώρα ο κύριος Γαοντινάζη. Από την Ουγγαρία παρακαλώ. Érdeklődéssel hallgatom a vitát, és elgondolkozom azon a aspektuson, amit a bizottság képviselője vetett föl, mégpedig azt, hogy valóban a demokratikus deficitet ért. Ευχαριστώ. Παρακολούθησα την συζήτηση και ο εκπρόσωπος της Επιτροπής μας είπε ότι πρέπει να μειώσουμε το δημοκρατικό έλλειμμα, ότι αξίζει τον κόπο. Για κάποιον δευματολόγο είναι ενδιαφέρον να ξέρει γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση αναλαμβάνει μια τέτοια δράση. Γιατί υπάρχουν παράλληλες διαδικασίες. Γιατί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει δικαίωμα πρωτοβουλίας. Γιατί δεν μπορεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να κάνει νομοθετική πρόταση. Οι ευρωβουλευτές εκλέγονται από τους Ευρωπαίους πολίτες με καθολική ψηφοφορία. Οπότε οι ευρωβουλευτές υποστηρίζουν τα συμφέροντα των διαφόρων χωρών που εκπροσωπούνται μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τα συμφέροντα αυτά πρέπει να ενισχύονται με μια νομοθετική πρόταση. Η συζήτηση παίρνει κακό δρόμο κατά τη γνώμη μου. Είναι σημαντικό να δίνουμε τη δυνατότητα στον κόσμο να συμμετέχουν στη δημοκρατία λέγοντας απευθείας τη γνώμη τους. Εδώ όμως όπως σας είπα παίρνουμε στραβό Υπάρχουν πολλές ρήτρε διασφάλισης μέσα στο κείμενο. Λέμε για παράδειγμα ότι άπαξ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θέλει να δώσει συνέχεια σε μία πρόταση, παρόλα αυτά να πρέπει να απαντήσει. Ή μιλάμε για τις ευρωπαϊκές αξίες, ότι αν δεν συνάδει με τις ευρωπαϊκές αξίες μια πρωτοβουλία, τότε απορρίπτεται. Ναι, αλλά ποιος το αποφασίζει αυτό. Αυτές είναι αυθαίρετες αποφάσεις. Σε μια δημοκρατία είμαστε αξιόπιστοι μόνο εφόσον οι βουλευτές, οι εκλεγμένοι δηλαδή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη συγκεκριμένη περίπτωση, να μπορούν να κάνουν ομοθετικές προτάσεις. Και να μην υπάρχει μονοπόλιο πρωτοβουλίας που στην συγκεκριμένη περίπτωση το έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βέβαια αυτή η συζήτηση έχει ξαναγίνει, είναι παλιά. Εδώ, αντί να τα βάλουμε με τις αιτίε, τα βάζουμε με τις συνέπειες. Νομίζω ότι αυτό το φιλτράρισμα που αναφέρεται στην πρόταση θα οδηγήσει σε ένα τεράστιο διοικητικό εμπόδιο για τους πολίτες. Τα ποσοστά, για παράδειγμα, που πρέπει να επιτευχθούν. Νομίζω ότι ο Ευρωπαίος πολίτης θα δυσκολευτεί πάρα πολύ για να φτάσει εκεί που πραγματικά γίνονται οι διαπραγματεύσεις μέσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και έτσι φοβάμαι ότι πολλά θέματα θα μείνουν απ' έξω. Στη χώρα μου για 40 χρόνια είχαμε δικτατορία. 40 χρόνια λοιπόν υπήρχε ένα μόνο κόμμα το οποίο έλεγε τι ήταν καλό και τι ήταν κακό. Αυτό αποφάσιζε. Ο δρόμος αυτός λοιπόν που έχουμε πάρει δεν είναι καλός ναι, να ενισχύσουμε την άμεση τη συμμετοχική δημοκρατία, ναι, να έχουμε στη διάθεσή μας ένα τέτοιο μέσο, όπως είναι η ΠΕΠ, που προβλέπεται εξάλλου από τη συνθήκη της Λισαβόνας, αλλά είναι πολύ σημαντικό οι ευρωβουλευτές να έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν προτάσεις πρωτοβουλίας, να λαμβάνουν την πρωτοβουλία δηλαδή για νομοθετικές προτάσεις. Πιστεύω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι εδώ για να υποστηρίζει τον κόσμο και όχι για να δημιουργήσει ένα υπερέθνος. Από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Thank you, Madam Chair. το Ελληνικό Κοινοβούλιο Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων συζήτησε αναλυτικά την πρόταση και βρίσκει ότι ε, είναι ισορροπημένη στα βασικά της χαρακτηριστικά και κυρίως είναι ισορροπημένη στις ε, τυπικές προϋποθέσεις οι οποίες πρέπει να πληρούνται για να τεθεί σε κίνηση η πρωτοβουλία των πολιτών. Υπάρχει όμως η εξής παρατήρηση. Το κείμενο της Επιτροπής α, τουλάχιστον στα μάτια ενός νομικού που είναι και πολιτικός α, έχει μια ουδετερότητα. Θα την έλεγα μια α, χρυσή ουδετερότητα, γραφειοκρατική ουδετερότητα, πάντως μια ουδετερότητα που δεν είναι βέβαιο ότι την συναντάμε συχνά στην κοινωνία. Τι θέλω να πω. Το, η πρόταση της Επιτροπής αναφέρεται σε μια πρωτοβουλία πολιτών η οποία θα ζητά από την Επιτροπή να παρέμβει, να θέσει σε κίνηση νομοθετική πρωτοβουλία για ρύθμιση ενός θέματος. Στην πραγματικότητα αυτό το οποίο πιθανότατα θα έχουμε είναι πρωτοβουλία πολιτών, όχι δίνοντας απεριόριστη διακριτική ευχαίρεια στην Επιτροπή για νομοθετική ρύθμιση θέματος, αλλά δίνοντας ή απαιτώντας συγκεκριμένη in concrete νομοθετική ρύθμιση. Με βάση, αν έχουμε αυτό το μοντέλο πρωτοβουλία πολιτών, υπάρχει το εξή για την Επιτροπή η Επιτροπή να, το πρώτο είναι η Επιτροπή να δεχθεί ότι η πρόταση είναι παραδεκτή, να βάλει μπροστά την διαδικασία, αλλά επί της ουσίας να προτείνει αντίθετα πράγματα από τα συγκεκριμένα που ζητάνε οι πολίτες. Και εδώ θα υπάρχει ένα θέμα. Η ΜΕΝ Επιτροπή θα χρησιμοποιεί την πρωτοβουλία των πολιτών για να καταλήξει σε ένα αποτέλεσμα το οποίο μπορεί να είναι διαφορετικό. Και εδώ πρέπει να το δούμε. Το δεύτερο ζήτημα το οποίο μας απασχόλησε είναι ότι στις γενικές αρχές, και αυτό είναι μέσα στο δικαιοδοτικό μας σύστημα, είναι πολύ γνωστό σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, συχνά οι γενικές αρχές επιτρέπουν μια καταχρηστική α, αξιολόγησή τους. Στην προκειμένη περίπτωση, το είπαν και άλλοι συνάδελφοι, μια καταχρηστική άρνηση της Επιτροπής να αποδεχθεί το παραδεκτό μιας πρότασης είναι ανέλεγκτη. Το ερώτημα είναι, δεν θα μπορούσε στα πλαίσια ενός συστήματος ελέγχου και ισορροπιών το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ελέγχει την Επιτροπή μέσα από συγκεκριμένη διαδικασία για, το, για την απόρριψη ενός αιτήματο πρωτοβουλία πολιτών. Και η τελευταία παρατήρηση, ότι μιας και μπαίνουμε όλο και ταχύτερα σε μια, σε μια εποχή με ηλεκτρονικές επικοινωνίες, γιατί η Επιτροπή δεν μπορεί να προσφέρει τον δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στον δικτυακό τόπο καλύτερα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μια συγκεκριμένη διεύθυνση στην οποία να καταχωρούνται όλες οι πρωτοβουλίες, να ενημερώνονται οι πολίτες μέσα από αυτή τη διεύθυνση και να μπορεί να γίνεται αυτή η ανταλλαγή των, και η συλλογή των υπογραφών, αλλά και η ενημέρωση ταυτόχρονα μέσα και με την υποστήριξη, την τεχνική υποστήριξη, την ηλεκτρονική υποστήριξη της Επιτροπής. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πολύ. Ο Επίτροπος είπε πριν ότι και οι πολίτες έχουν να κερδίσουν από όλη αυτή τη διαδικασία που προβλέπεται από τη συνθήκη της Λισαβόνας. Η πρωτοβουλία Ευρωπαίων πολιτών όμως σε μένα μου δημιουργεί κάποιες αμφιβολίες αν όντως από αυτήν έχουν τελικά να κερδίσουν. Διότι Εμάς μας ενδιαφέρει όχι μόνο οργανωμένες, οργανώσεις, συνδικάτα και τα λοιπά να μπορούν να αναλάβουν μια τέτοια πρωτοβουλία, αλλά να μπορούν να αναλάβουν τέτοια πρωτοβουλία και απλοί πολίτες. Και για αυτούς να είναι εύκολο στην πράξη να υποβάλουν μια τέτοια πρωτοβουλία η οποία θα καταλήξει και κάπου. Λέτε το 1 τρίτο των χωρών μελών πρέπει να εκπροσωπείται για μια τέτοια πρωτοβουλία. Εδώ το είδατε, υπάρχουν διαφορετικές προτάσεις για τον αριθμό των χωρών. Λέμε ότι θέλουμε να είναι λιγότερες, να είναι το 1 τέταρτο και το 1 πέμπτο μάλιστα των χωρών που να φτάνει. 1 τέταρτο τουλάχιστον. Οι περισσότεροι νομίζω εδώ μέσα συμφωνούν για να είναι το 1 τέταρτο, αν όχι και λιγότερες χώρες. Έπειτα υπάρχει ο κίνδυνος για υπερβολική γραφειοκρατία για την επαλήθευση των υπογραφών που έχουν συγκεντρωθεί ή υπάρχει το ζήτημα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των ανθρώπων που υπογράφουν ή το θέμα της πρωτοβουλίας προκειμένου αυτή να συνάδει με τις ευρωπαϊκές αξίες, ότι πρέπει να υπάρξει ένας κώδικας που θα οδηγήσει φοβάμαι σε ένα ταμπού. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να αποφύγει τέτοιου είδου πρωτοβουλίε. Εγώ διαβάζω μερικά άρθρα ορισμένων από τη δεξιά που λένε ότι μήπως υπάρξει κάποια πρωτοβουλία για τον περιορισμό της μετανάστευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή ότι δεν θα πρέπει να δεχτούμε, λένε άλλοι, κάτι σχετικά με την προσχώρηση της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή υπάρχουν και πράγματα που δεν έχουν άμεσα να κάνουν με την αξίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέτοιου είδους θέματα καταλήγουν να γίνονται ταμπού. Και πολύ εύκολα φοβάμαι ότι μπορεί να διηγηθούμε σε λαϊκισμό και να καταπνίγεται κάθε πρωτοβουλία ήδη από την αρχή. Για τους ελέγχους τώρα. Υπάρχει πρόταση του Κοινοβουλίου στην οποία βλέπω ότι θέλουμε να ελέγχεται η ιδεολογία, το κατά πόσο δηλαδή συνάδει με τις ευρωπαϊκές αξίες ή όχι μια πρωτοβουλία, ήδη από την αρχή. Εγώ δεν το βλέπω αυτό στο κείμενο της Επιτροπής, γιατί εκεί λέει ότι πρέπει να έχουν μαζευτεί 300.000 υπογραφές, μπορεί τελικά να καταλήξουμε στο να είναι 100.000, δεν ξέρω, αλλά τελικά τι θα γίνει, θα υπάρξει πρώτα η επαλήθευση τη τιμή της καταχώρησης, μια πρωτοβουλία κατά πόσο συνάδει με τι ευρωπαϊκέ ε, αξίε ή τέλο πάντων με τις αρμοδιότητες Ευρωπαϊκή Επιτροπής ή αργότερα. Μήπως μπορούμε να έχουμε δύο διαφορετικά στάδια, δηλαδή στο πρώτο στάδιο με την καταχώρηση να ελέγχουμε κατά πόσο είναι σοβαρή και το πάντων συνάδει με τις ε, ε, ευρωπαϊκές αξίες και μετά αργότερα να δούμε για τα άλλα κριτήρια. Η συλλογή υπογραφών συγκεντρώνεται και τη στιγμή που θα πρέπει να αποφασίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τότε θα έχει σταματήσει αυτή η συλλογή μέχρι να πάρει την αποφασή της Επιτροπή και μετά θα συνεχίζεται η συλλογή, έτσι δεν είναι. Θα ήθελα να μου διευκρινίσετε περισσότερο τι θα γίνει με αυτές τις περιπτώσεις. Ζήτω συγγνώμη, αλλά θα πρέπει να απουσιάσω από εδώ και πέρα γιατί δυστυχώς έχω κάποιες άλλες δραστηριότητες και θα ήθελα να ζητήσω από τη φίλη Τσίτα Γκορμάη να πάρει τη θέση μου. Θα ήθελα να χαιρετήσω εκ νέου τον Επίτροπο Σεύκοβιτς, την εκπρόσωπο της Βελγικής Βουλής και τη συμπρόεδρο αυτής εδώ της συνάντησης, την κυρία Ματσόνη, προς την οποία θα ήθελα να ζητήσω στο τέλος της συζήτησης να παρουσιάσει κάποια πρώτα συμπεράσματα. Σας ευχαριστώ προσωπικά, σας χαιρετώ. Ευχαριστώ κύριο Στυλιανίδης. Έχει το λόγο τώρα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχω την πεποίθηση ότι αυτή η μεγάλη αλλαγή που έρχεται από τη συνθήκη της Λισαβόνας όσο και αν καμιά φορά θέλουμε να το κρύψουμε είναι μια κίνηση ακροβάτη σε τεντωμένο σχοινί. Απ' τη μια όντως δημιουργεί προϋποθέσεις να περιοριστεί το δημοκρατικό έλλειμμα να νιώσει ο πολίτης, ο Ευρωπαίος πολίτης ότι έχει λόγο στους θεσμούς αλλά από την άλλη υπάρχει μεγάλο ενδεχόμενο εάν δεν προσέξουμε τις διαδικασίες να γελιοποιήσουμε την ίδια την πρωτοβουλία και να δημιουργήσουμε απεριόριστα προβλήματα στο θεσμικό οικοδόμημα Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήδη έχουν υποθεί πολλά γύρω από κάποιες αντιφάσεις που εμφανίζονται στην έννοια του παραδεχτού και στο γεγονός ότι υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να απογοητεύσουμε τους πολίτες πριν ακόμη ξεκινήσουν. Εμείς ως Κοινοβούλιο της Κύπρου Έχουμε συζητήσει εκτεταμένα. Ήδη έχουμε στείλει και είναι μπροστά σε όλους σας οι γενικές μας θέσεις με, διάφορες, με διαφοροποιήσεις κομμάτων. Είμαστε θετικοί στις προτάσεις. Έχουμε κάνει και κάποιες πιο εξειδικευμένε προτάσεις. Αλλά θέλουμε να επισημάνουμε αυτό. Ότι όταν θα ξεκινήσει αυτή η πολύ μεγάλη τομή θα πρέπει να είμαστε απολύτως σίγουροι και έτοιμοι ότι η κίνηση του ακροβάτη θα καταλήξει στο τέρμα. Θα επισημάνω δύο παρατηρήσεις μόνο, οι οποίες είναι πάρα πολύ σημαντικές. Όντως, είναι αδιανόητο η Επιτροπή να είναι και ο ελέγχο και ο ελεγχόμενος. Αυτό πρέπει εξ αρχής να αποκλειστεί γιατί μιλούμε για δημοκρατική αντίφαση εκ προημίου. Το δεύτερο, και παραμένω στο θέμα του παραδεχτού γιατί θεωρώ τα υπόλοιπα είναι ίσως σε κάποιο σημείο δευτερεύοντα, εάν θα αποδεχτούμε την πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για μια επιτροπή σοφών να αξιολογεί το θέμα του παραδεχτού ημί, θα πρέπει να γίνεται όσο το δυνατό πιο σύντομα στη διαδικασία αλλιώς θα δημιουργηθεί η εικόνα στους Ευρωπαίους πολίτες ότι υπάρχει ένα φιλτράρισμα εκ των άνω που ουσιαστικά τους απαγορεύει να μπουν ίδιοι, να γίνουν μέρος των θεσμών οι ίδιοι και της θεσμικής διαδικασίας. Ευχαριστώ. Ehm, Ευχαριστώ πολύ. Η Κοινοβούλιο της ε, Εστονία τώρα. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, το Εστονικό Κοινοβούλιο έχει συζητήσει επίσης την Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών. Το κάναμε αυτό και φέτος αλλά ήδη τον Ιανουάριο και η κυβέρνηση της Εστονίας ε, συζήτησε πάνω σε αυτό. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης μας μάλιστα γνωμοδότησε και εγώ η ίδια εκπροσώπησα τους πρασίνους, αλλά δεν προσκλήθηκα στην συζήτηση. Άρα το δικό μου πολιτικό κόμμα μπορώ να πω ότι δεν συμφωνεί με όλα όσα αποφασίστηκαν στην Εστονία. Και δεν μπορώ εγώ προσωπικά να συμφωνήσω με όλα όσα συμπεριλαμβάνονται στην επίσημη θέση της Εστονίας. Πάντως, θέλω να προσθέσω κάτι το οποίο δεν έχουμε ακούσει ακόμα. Το Κοινοβούλιο της Εστονίας έστειλε επιστολή στην Επιτροπή και είπε ότι εμείς στηρίζουμε ειδικέ προϋποθέσεις για όσους προτείνουν Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία, όπου να φαίνεται ποιος μπορεί να υποβάλει τέτοια πρωτοβουλία και να ελέγχεται η αξιοπιστία του ατόμου ή των ατόμων που υποβάλλουν πρωτοβουλία Ευρωπαίων πολιτών. Ότι πρέπει επίσης να φαίνεται πώς χρηματοδοτείται ο διοργανωτής μιας τέτοιας πρωτοβουλίας. Όσον αφορά τώρα τις υπογραφές και τον αριθμό των υπογραφών, η κυβέρνηση της Εστονής πιστεύει ότι έξι μήνες φτάνουν για να συγκεντρωθούν όλες οι το κόμμα μου όμως δεν συμφωνεί με μια τέτοια προθεσμία γιατί δεν τη βρίσκουμε ρεαλιστική. Η Επιτροπή Σταγματικών ε, Υποθέσεων στο Κοινοβούλιο μας αποφάσισε να συζητηθεί το θέμα στην Επιτροπή Ευρωπαϊκών Θεμάτων. Και η Επιτροπή Ευρωπαϊκών Θεμάτων του Ιστονικού Κοινοβουλίου είπε ότι δεν πρέπει να συμφωνήσουμε με ένα τρίτο ή ένα τέταρτο των χωρών μελών αλλά πιστεύουμε ότι πρέπει να είναι πολίτες από περισσότερες χώρες. Οπότε στην Εστονία πρέπει να ξαναρχίσει η συζήτηση γιατί πολλά από τα θέματα είναι επίμαχα ακόμα. Θα ήθελα ε, κυρία Ρίτεν, θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συμμετέχοντες στη συζήτηση αυτή. Θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί όπως είπαμε και στην αρχή πρόκειται εδώ πέρα για κάτι πολύ ειδικό. Έχω ακούσει λοιπόν τόσους εκπροσώπους τόσο από το Αθηνικά Κοινοβούλιο όσο και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πιστεύω ότι υπάρχει μια βάση για τη συζήτηση και είναι το τι συμπεριλαμβάνεται στην συνθήκη. Εκεί υπάρχει ένα εκατομμύριο πολίτες λέει επίσης από ένα σημαντικό αριθμό χωρών μελών η συνθήκη και λέει επίσης στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι τρία στοιχεία τα οποία προβλέπονται ήδη από τη συνθήκη της Λισαβόνας. Οπότε αυτό είναι το σημείο κίνηση για να προχωρήσουμε και να καταλήξουμε σε ένα κανονισμό. Τώρα τα άλλα όρια είναι πράγματα τα οποία μπορούμε να τα συζητήσουμε. Και ακριβώ ακούσαμε κριτική από πολλούς από εσά επειδή δεν είναι κάτι που προβλέπεται από τη συνθήκη. Αναφέρονται, λοιπόν, όπως είπαμε, κάποια όρια στην ε, συνθήκη και αυτό. Γιατί όπως καταλαβαίνετε η πρωτοβουλία Ευρωπαίων πολιτών είναι ένα σοβαρό θέμα, είναι ένα σοβαρός μηχανισμός που κοστίζει και δεν μπορούμε να διαφορήσουμε εντελώ. Δεν μπορεί δηλαδή κάποιο να χρησιμοποιεί αυτό τον μηχανισμό για το τίποτα, για ψηλουπίδημα. Δεν είναι και αυτός ο στόχος του μηχανισμού. Είναι ένας μοναδικός μηχανισμός από τη φύση του, του οποίου τα αποτελέσματα θα πρέπει να οδηγήσουν σε μια νομοθετική πρόταση κανονικά. Ξέρω και από το Βέλγικο Κοινοβούλιο, όπου έχουμε συζητήσει κάπως, αλλά έχουμε ξεκινήσει αργά και πρέπει να συζητήσουμε ακόμα. Τώρα κάποιες παρατηρήσεις για αυτά που άκουσα εδώ. Αυτά που είπατε για τη γραφειοκρατία, συμφωνώ, όντω είναι κάτι που επιβαρύνει πολλές φορές στις διαδικασίες, το είπαν ε, όλες οι χώρες, παντού ισχύει, δεν θέλουμε να βαρύνουμε τη διαδικασία με γραφειοκρατία. Επίσης, να χρησιμοποιήσουμε όσο γίνεται περισσότερο τη σύγχρονη τεχνολογία. Το είπε και ο Επίτροπο. Η Ευρώπη πρέπει να είναι μια Ευρώπη του μέλλοντο. Δεν έχει νόημα να κοιτάμε προ τα πίσω. Όχι, πρέπει να χρησιμοποιούμε ό,τι τεχνολογία έχουμε στη διάθεσή μα. Και γι' αυτό και εγώ ε, συμφωνώ. Επίση, να βοηθήσουμε να συμμετέχουν όσο γίνεται περισσότερο οι νέοι. Η ηλικία των 16 είναι όντω μία δυνατότητα. Μπορεί κανεί βέβαια και να αναρωτηθεί γιατί να υπάρχει όριο ηλικία. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, συμφωνώ και εγώ με τον προβληματισμό σα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλε σα τι παρατηρήσει. En uh, men meldt mij dat er nog een collega is uit uh, Polen, het Poolse parlement, meneer. Ο κύριο Κίκο από το Πολωνικό Κοινοβούλιο. Έχετε το λόγο. Κοιτάξτε, όσον αφορά στο θέμα της ε, νομοθετικής πρωτοβουλίας ε, για τους Ευρωπαίους πολίτες, θα ήθελα να κάνω μία ερώτηση. Ένα εκατομμύριο άνθρωποι μπορούν να έχουν μεγαλύτερη εξουσία από τους ε, ερετούς εκπροσώπους των πολιτών, από τους βουλευτές. Γιατί σε αυτή τη φάση η νομοθετική ρύθμιση είναι παράλογη. Το Κοινοβούλιο έχει περιορισμένες εξουσίες σε σύγκριση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μπορούμε να πούμε ότι από πλευρά, σε επίπεδο εξουσίας, εκτός από τις αρμοδιότητες στον προϋπολογισμό, οι νομοθετικές αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι αμελητές, αν τις συγκρίνει κανείς με αυτές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Γι' αυτό λοιπόν, αν χρησιμοποιήσουμε την πρωτοβουλία των πολιτών ως ένα μέσο για να θεσπίσουμε νόμους και μετά να αφήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποφασίσει κατά πόσον θα αναλάβει πρωτοβουλίες με βάση την πρωτοβουλία των πολιτών, μήπως με τον τρόπο αυτό πέφτουμε στην παγίδα όπου τελικά ε, τις αποφάσεις λαμβάνει αποκλειστικά και μόνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα είναι εκείνη που θα αποφασίζει κατά πόσον μια πρωτοβουλία συμβαδίζει όχι με τις ευρωπαϊκές αξίες και κατά πόσον εντάσσεται στις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ λοιπόν πιστεύω ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με έλλειψη νομιμότητας, νομοποίησης απέναντι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γιατί το Κοινοβούλιο είναι εκείνο που εκλέγεται άμεσα και πρέπει να έχει περισσότερες νομοθετικές αρμοδιότητες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το επόμενο θέμα έχει σχέση με το όριο ηλικία ε, το να μετατεθεί προς τα κάτω. Είμαι κατά του να πάει στα 16 χρόνια, ετέθη το ερώτημα κατά πόσον θα πρέπει να εισαχθεί ή όχι όριο ηλικία. Αυτό δηλαδή μήπως ε, σημαίνει ότι θα πρέπει και τα παιδιά 13 ετών να υπογράφουν την πρωτοβουλία. Αν δεν υπάρχει όριο ηλικία, τότε ε, να μπορεί να υπογράφει καθένας, οποιαδήποτε ηλικία και αν βρίσκεται. το όριο ηλικία έχει σχέση και με την ε, ψυχολογική οριμότητα ενός ανθρώπου για να αποφασίσει. Και έχει σχέση και με την κοινωνικοποίησή του, με την ανατροφή των παιδιών. Είναι λοιπόν απόλυτα φυσιολογικό να θεωρούμε ότι σε ηλικία 18 ετών μπορεί ένας άνθρωπος να λάβει αποφάσεις και ε, πολύ πιο δύσκολα γίνεται αντικείμενο δόλιων χειρισμών. Ενώ ο μικρότερος είναι πολύ πιο ευάλωτος και πολύ, μπορεί πολύ πιο εύκολα να επηρεαστεί από τα πολιτικά κόμματα. Οι νέοι κατά κανόνα είναι πολύ παρορμητικοί και ως εκ τούτου πολύ εύκολα μπορούν να πέσουν θύματα σε αξίες που δεν έχουν ε, και μεγάλη σημασία. Νομίζω έχουμε άλλη μισή ώρα περίπου. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να δώσω το λόγο ε, στον κύριο Σέφοβιτς, ε, μετά θα ζητήσουμε τον κύριο Ρότ να κάνει τα σχόλια και κατόπιν οι συγητές. Και τέλος έχουμε την πρόεδρο της Επιτροπής Αναφορών η οποία θα πάρει τα πέντε της ε, λεπτά πριν ε, κάνουμε τις ε, καταληκτικές παρατηρήσεις. Αυτά για το χρονοδιάγραμμα. Αν μου επιτρέπετε λοιπόν θα ήθελα να δώσω το λόγο στον αντιπρόεδρό μας που ασχολείται πολύ με τα θέματα αυτά και μπορώ να πω ε, στον Πολωνό συνάδελφο ότι κοιτάξτε δουλεύουμε πολύ σκληρά για να βρούμε μια ε, ισόρροπη απάντηση. Ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να έχει φωνή και προσπαθούμε να δούμε πώς μπορεί να επικρατήσει η ισορροπία. Ευχαριστώ Ζήτα. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω την κυρία Ρούτε από το Βέλγιο που μας υπενθύμησε ποιες ακριβώς είναι οι παράμετροι που περιχαρακώνουν την πρωτοβουλία. Ένα εκατομμύριο λοιπόν υπογραφές που να έρχονται από διάφορα κράτη-μέλη και η πρωτοβουλία μπορεί να απευθύνεται στην Επιτροπή μόνο εφόσον η Επιτροπή έχει δικαίωμα νομοθεσίας ε, σε αυτόν τον συγκεκριμένο τομέα για τον οποίο γίνεται λόγος. Οτιδήποτε άλλο, ε, δε, για οτιδήποτε άλλο δεν μπορεί να αναλυφθεί πρωτοβουλία ε, πολιτών. Και δεν έχει νόημα να υποσχεθεί κανείς κάτι τέτοιο στους πολίτες, γιατί οι Κομισιόν ε, υπάρχουν και τομείς οι οποίους δεν μπορεί να νομοθετήσει, πέρα από αυτούς που τους έχουν ανατεθεί. Ε, την πρώτη ερώτηση για το οικονομικό βάρος και για τη διαδικασία επαλήθευσης. Νομίζω εδώ αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε είναι ε, να βρούμε ε, τις ε, πιο φιλικές προς το χρήστη λύσεις. Λέμε λοιπόν ότι εναπόκειται στους ίδιους τους πολίτες να αποφασίσουν μόνοι τους το πώς θα επαληθεύουν τις υπογραφές. Για την Επιτροπή δεν έχει καμία απολύτως σημασία πώς θα γίνουν όλα αυτά. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς προτείνουμε ότι για μας είναι απόλυτα εντάξει ε, τα κρατημέλη να προβαίνουν σε δειγματοληπτικούς ελέγχους ε, για να διαπιστώσουν ε, κατά πόσον οι υπογραφές είναι γνήσιες ή όχι. Πάντως πρέπει να υπάρχει κάποιος έλεγχος και αυτός ε, αν γίνεται από τα κράτη-μέλη, ο έλεγχος αυτός ε, θα είναι και πολύ, πιο εύκολος. Τώρα, να ερωτήθηκαν και κάποια άλλα, τέσσερα κάποια άλλα ερωτήματα σχετικά με το τι είναι επιτρεπτό. Ε, στις εισαγωγικές μου παρατηρήσεις νομίζω εξήγησα πόσο σημαντικό είναι Ε, θα ήθελα λοιπόν ε, να δεχθώ τα σχόλια των Μπόνος και Καλτανάκη. Ποιος είναι τελικά εκείνος που αποφασίζει. Ποιε είναι οι Ευρωπαϊκέ αξίε, ποιε είναι οι σοβιετικέ αξίε. Εγώ σπούδασα στη Σοβιετική Ένωση και πρέπει να σα πω ότι οι ευρωπαϊκές αξίες διαφέρουν πάρα πολύ από τι Σοβιετικέ και νομίζω μπορούμε να κάνουμε αυτή τη διάκριση. Νομίζω ότι περισσότεροι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εύκολα μπορούν να κάνουν το διαχωρισμό ανάμεσα σε ευρωπαϊκέ και σοβιετικές αξίε. Και αν υπάρχουν και αμφιβολίες έχουμε ε, τον χάρτη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πολλά άλλα σχετικά έγγραφα. Ε, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να είναι κανείς πυρηνικός φυσικός για να αποφασίσει και να καταλάβει τι είναι ευρωπαϊκό και τι είναι αντιευρωπαϊκό. Εν πάση περιπτώσει, αν παρόλα αυτά εξακολουθούν να υπάρχουν αμφιβολίες και αν η Κομισιόν κάνει κατάχρηση της θέσης της, ε, τότε θα υπάρχει η δυνατότητα προσφυγής προσβολής της απόφασης στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο όπως και με οποιαδήποτε άλλη απόφαση που λαμβάνει η Κομισιόν. Νομίζω λοιπόν ότι εδώ έχουμε αδιάσυστα στοιχεία και έλεγχο για ε, να ξεκινήσουμε πριν δρομολογηθεί η πρωτοβουλία των πολιτών. Όσον αφορά στο θέμα που έθεξε ο κύριος Αλευράς από την Ελλάδα. Ο κύριος Λαμασούρ νομίζω κατέστησε απόλυτα σαφές ότι σε αυτό το συγκεκριμένο θέμα η Επιτροπή ε, θα συμπεριφέρεται σαν να έπαιρνε ένα νομοθετικό ψήφισμα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γιατί πρέπει την πρωτοβουλία να την κρίνουμε και ως σημαντική αλλά και ως πρωτοβουλία που καθορίζει την ατζέντα. Άρα δηλαδή η Κομισιόν πρέπει να μπορεί να διαφυλάσει το δικαίωμά τη ε, να αναλαμβάνει την πρωτοβουλία. Ακούει βέβαια την άποψη των πολιτών, αλλά επειδή πρέπει να σεβόμαστε του θεσμού και τη θεσμική ισορροπία, πρέπει και να σεβόμαστε ότι η Κομισιόν είναι εκείνη που έχει το δικαίωμα πρωτοβουλία και να πρόκειται στην Κομισιόν να αποφασίσει αν θα νομοθετήσει εφόσον το ζητούν οι πολίτε ή αν δεν θα νομοθετήσει καθόλου. Γιατί μπορούμε να έχουμε πρωτοβουλίες πολιτών που ε, μπορεί να συγκεντρωθούν ε, ε, υπογραφές, αλλά το θέμα δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Κομισιόν και εκεί δεν μπορεί να νομοθετήσει. Ας πούμε για τα περιβαλλοντικά ή για την γονική άδεια, του να περιστεί η γονική άδεια ή να καταργηθεί. Αυτό δεν είναι... Αυτό είναι η αρμοδιότητα της Κομισιόν, αλλά η απόφαση θα ήταν αρνητική. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να καταργηθει αυτο δεν ειναι αυτο ειναι σε αρμοδιοτητα της κομισιον αλλα η κατά νου ότι η Κομισιόν έχει ε, νομοθετικό μονοπόλιο. Η Κομισιόν θα είναι ο σημαντικότερος παίκτη ε, και ο μόνος νομοθέτης. Η απάντηση είναι όχι, γιατί εμείς έχουμε μόνο το δικαίωμα να καταθέσουμε πρόταση. Και μετά βέβαια θα προκύψει συζήτηση όπως αυτή που έγινε σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, δηλαδή ε, ανάμεσα στα κράτη-μέλη ε, εκεί θα αποφασιστεί κατά πόσον στηρίζουν την νομοθετική πρόταση. Γιατί εμείς καταθέτουμε την πρόταση, αλλά νομοθέτες είναι ε, το ε, Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εφόσον η πρόταση φτάσει και μέχρι τη φάση της νομοθεσίας. Τώρα, αυτά που είπε ο κύριος Κλάς από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ο κύριος Τηλιανίδης σχετικά με την προστασία των δεδομένων. Και πάλι λοιπόν εδώ προσπαθήσαμε να βρούμε τη βέλτιστη δυνατή λύση. Γιατί νομίζω ότι βεβαίως και όλοι συμφωνούμε ότι είναι απαραίτητο να συμπεριλάβουμε την ε, online συγκέντρωση των υπογραφών γιατί αλλιώ ε, το σύστημα θα είναι απαρχαιωμένο. Από τη στιγμή λοιπόν που το δέχεται κανείς αυτό προφανώς και παρισφρύνουν σημαντικές ανησυχίες σε σχέση με την προστασία των ε, προσωπικών δεδομένων. Πολύ ευαίσθητο θέμα. Ξέρετε ότι σήμερα μπορεί να γίνουν δόλοι χειρισμοί, καταχρήσεις πρέπει να είμαστε προσεκτικοί για το πώς ε, θα προτείνουμε να ε, την χάνουν, ποιον χειρισμών θα πρέπει την χάνουν ε, τα δεδομένα, πώς θα προστατεύονται. Εμείς θέλουμε να εφαρμόσουμε όλα τα ευρωπαϊκά στάνταρτ σε αυτό το θέμα. Και οι οργανωτές και αυτοί να φέρουν ευθύνη για την προστασία των δεδομένων. Γιατί αυτοί που συγκεντρώνουν τις υπογραφές είναι και υπεύθυνοι για την προστασία τους. Εδώ λοιπόν και πάλι σεβόμαστε ε, την εθνική νομοθεσία. Σε μια χώρα, ας πούμε, η προστασία υπόκειται στο αστικό δίκαιο. Σε άλλη χώρα, η προστασία των δεδομένων υπάγεται στο ποινικό δίκαιο. Εναπόκειται λοιπόν ε, στο εκάστοτε κράτος μέλος και στη νομοθεσία του για το πώς ε, θα χειρίζεται το θέμα αυτό. Βεβαίως η προστασία αδιαμφισβήτητα είναι σημαντική. Όσον αφορά τη συνάδελφο από την Εστονία, πληροφορίες σχετικά με τους οργανωτές. Γιατί το συμπεριλάβαμε αυτό διότι πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό για τη διαφάνεια. Είναι ε, ένα απλό ερωτηματολόγιο που αναφέρει κανείς ποιος είναι ο οργανωτής, ποιος είναι ο στόχος της πρωτοβουλίας και βεβαίως ε, πώς ε, χρηματοδοτούνται οι πρωτοβουλίες. Γιατί νομίζω ότι ο κύριος Κλάς είπε ότι δεν θα ήθελε να υπάρχει ένα εργαλείο το οποίο να το χρησιμοποιούν μόνο τα οργανωμένα πολιτικά κόμματα, οι μεγάλες μικαιότητα, συνδικάτα. Αν θέλουμε λοιπόν η κατάσταση να είναι απόλυτα σαφής ότι αυτό είναι το εργαλείο για τους πολίτες, τότε πρέπει να εισάγουμε το στοιχείο της διαφάνειας, να γνωρίζουμε ποιοι είναι οι οργανωτές και ποιος χρηματοδοτεί. Γιατί θέλουμε να είμαστε σίγουροι ότι πίσω από τους οργανωτές δεν ε, κρύβονται κάποιες ομάδες πίεσης. Και από τη στιγμή που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε ένα τόσο σημαντικό δημοκρατικό εργαλείο για τις συζητήσεις μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει και να είμαστε απόλυτα σίγουροι ότι γίνεται σεβαστή η διαφάνεια και ότι ε, έχουμε στη διάθεσή μας όλα τα απαραίτητα δεδομένα για να έχουμε και μία σαφή εικόνα του ποιος είναι ο στόχος της πρωτοβουλίας και ποιοι είναι οι οργανωτές. Όσον αφορά στην ηλικία, απευθύνομαι στον συνάδελφο από την Πολωνία. Βλέπω ότι έχετε έντονη συζήτηση, διάσταση απόψεων. Εσείς λέτε ότι είστε κατά του να μειωθεί ε, το όριο, γιατί... Ε, μάλλον, Εσεί είστε υπέρ του να μειωθεί. Υπάρχουν όμω και άλλοι που λένε ότι όχι, να σεβόμαστε το όριο που προβλέπεται στο νόμο. Είναι σαφές ότι η επαλήθευση είναι πολύ πιο εύκολο να γίνει με, εφόσον έχουμε εκείνους ε, που βρίσκονται σε ηλικία ε, που έχουν δικαίωμα ψήφου και έχουν καταγραφεί στα εκλογικά μητρώα. 16 βέβαια είναι στην Αυστρία και 18 ε, στα υπόλοιπα κρατημέλη αυτή η ηλικία. Πάντως είναι ένα από τα θέματα τα οποία θα συζητήσουμε ε, στην επόμενη τριμερή συζήτηση. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα δώσω το λόγο τώρα στον κύριο Βότ για τις τελικές του παρατηρήσεις. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει κάποια διάσταση απόψεων και εγώ θα ήθελα να τοποθετηθώ σε αυτήν. Πρώτον, όσον αφορά τον ελάχιστο αριθμό των κρατών μελών. Εδώ θα ήθελα να παρακαλέσω να εξετάσουμε το ενδεχόμενο να μειωθεί το όριο ηλικίας. Επισημάναμε τις, ε, τα κρατικά προσκόμματα και νομίζω ότι μπορούμε να μιλήσουμε για δημοκρατική πρωτοβουλία μόνο εφόσον ε, την πρωτοβουλία αυτή την ασπαστούν η πλειοψηφία των πολιτών των κρατών μελών. Είναι εξάλλου σημαντικό να έχουμε και ένα σημαντικό αριθμό ε, κρατών μελών αλλά επίσης θα πρέπει να έχουμε και όσο δυνατόν περισσότερους που να συμμετέχουν. Εγώ δεν θέλω να τα περιπλέξω περαιτέρω τα πράγματα. Και κάτι άλλο. Η έρευνα περί παραδεκτού να γίνεται στην αρχή. Γιατί διαπιστώθηκε ε, ότι η απογοητεύση είναι πολύ μεγάλη αν ε, σε κάποια μεταγενέστερη στιγμή αποφασιστεί τελικά ότι η πρωτοβουλία θα αποτύχει επειδή δεν βασίζεται στις προϋποθέσεις της συνθήκης της Λισαβόνας. Εκείνο το οποίο επίσης επιθυμώ είναι ε, η απόφαση της Κομισιόν να ελέγχεται σε τελευταίο στάδιο από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Αυτό το στοιχείο της ε, νομιμότητας ε, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο είναι το σωστό ανώτατο όριο προέκυψε κάποια διαφωνία στο θέμα του, ε, της κατώτερης ηλικίας, του ορίου ηλικίας. Το θέμα αυτό, γιατί δεν το αφήνουμε στα κράτη-μέλη. Σε κάποιες χώρες μπορεί κανείς να ψηφίσει σε ηλικία 16 ετών. Στις περισσότερες με τα 18 ή στα 21. Εγώ λοιπόν νομίζω ότι πρέπει να ε, προσαρμοστούμε στις εκάστοτε εθνικές παραδόσεις χωρίς να υπονομεύουμε την ευρωπαϊκή σημασία της πρωτοβουλίας. Και τέλος, αυτό που θέλω να καταστήσω σαφές είναι ότι αν τελικά η πρωτοβουλία στεφθεί από επιτυχία, χρειαζόμαστε και ε, κάποια δεσμευτικότητα. Κατά την άποψή μου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να λέει ότι έχει το μονοπόλιο πρωτοβουλίας. Θα πρέπει τουλάχιστον όσους αναλαμβάνουν και στηρίζουν την πρωτοβουλία σε αυτούς να εξηγεί τι ακριβώς θα γίνει με την πρωτοβουλία αυτή. Και έτσι η Κομισιόν οφείλει να συμπεριλαμβάνει και τα άλλα όργανα, άρα δηλαδή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ε, από εκεί ε, απορρέει ε, το γεγονός, το συμπέρασμα ότι η Κομισιόν είναι υπόλογη απέναντι στα άλλα όργανα. Ε, δεν ξέρω αν ο πίτροπος ή οι άλλοι το είπαν, αλλά, εν πάση περιπτώσει, ε, η συνθήκη της Λισαβόνας ισχύει εδώ και πάνω από ένα χρόνο. Εδώ και μήνες συζητάμε για την εφαρμογή ενός σημαντικού στοιχείου της συνθήκης της Λισαβόνας. Τώρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να εξετάσουμε προσεκτικά το θέμα, να δώσουμε χρόνο στον εαυτό μας, αλλά να μην ε, καθυστερούμε χωρίς λόγο. Ε, οι πολίτες οφείλουν ε, να κατανοήσουν και αυτοί ότι η πρωτοβουλία θα τεθεί σε ισχύ το συντομότερο δυνατόν. some questions concerning the Council, so I kindly ask him to, to react on. Merci, Madame la Présidente. Ο Σαστέλ λοιπόν, σημαντικό πρόσωπο λέει, πρόεδρος θα πάρει το λόγο. Καταρχάς ζητώ συγγνώμη από το, για, την, ε, κυρία, για τον κύριο Υπουργό ο οποίος αναγκάστηκε να φύγει. Ο κύριος Σεφκόβιτς απάντησε με μεγάλη ικανότητα στις περισσότερες από τις ερωτήσεις και δεν θα ήθελα να επανέλθω σε λεπτομέρειες. Υπήρχε ίσως ένα σημείο επί του οποίου θα πρέπει να σταθώ λίγο γιατί αφορά τα ίδια τα κράτη-μέλη. Είναι το θέμα της επαλήθευσης των προσωπικών δεδομένων, του ελέγχου των προσωπικών δεδομένων. Αρκετοί σταθήκατε στο θέμα αυτό και είπατε ότι θα πρέπει να αποφύγουμε βέβαια την γραφειοκρατία, την υπερβολική και θα βρούμε ένα σύστημα πρακτικό και μη γραφειοκρατικό. Αυτή είναι μια ανησυχία την οποία συμμερίζεται το Συμβούλιο και όπως είπε ο κύριος Επίτροπος θα προσπαθήσουμε να βρούμε ένα σύστημα ελέγχου στοιχείων προσωπικών το οποίο να είναι το πλέον ευέλικτο. Ταυτόχρονα θα ήθελα να θυμίσω ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ευθύνη στα κράτη-μέλη εδώ. Γιατί τα κράτη-μέλη σύμφωνα με τον κανονισμό θα είναι επιφορτισμένα να ελέγξουν τα δεδομένα αυτά. Και θα συμφωνήσετε μαζί μου λέγοντας ε, πως αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία γιατί θα πρέπει να δώσουμε εγγυήσει ε, στο σύστημα αυτό και στην αξιοπιστία του. Συνεπώς ο έλεγχος θα πρέπει να είναι σοβαρός. Θα πρέπει να είναι σοβαρός ο έλεγχος, πόσο μάλλον που ο έλεγχος αυτός θα πρέπει να γίνεται και με αρκετά μεγάλη ταχύτητα για να μην προκαλούνται καθυστερήσεις. Τρεις μήνες προβλέπει το σχέδιο του Συμβουλίου για τον έλεγχο των στοιχείων. Στα πλαίσια λοιπόν αυτής της λογικής, στην πρόταση του Συμβουλίου έχουμε προετοιμάσει ένα παράρτημα το οποίο προβλέπει ότι αναχώρα και ανάλογα με τα ειδικά εθνικά χαρακτηριστικά, νομικά εννοούμε, προβλέπεται να ελεγχθούν ε, μια σειρά δεδομένων κατά περίπτωση. Φυσικά το σύστημα αυτό θα πρέπει να είναι σε εισαγωγικά ελαφρύ, αλλά από την άλλη θα πρέπει να κατανοήσετε ότι για τα κράτη-μέλη το θέμα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η συζήτηση που προηγήθηκε μπορώ να σας πω ότι δεν ήταν ιδιαίτερα εύκολη και θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ισπανική Προεδρία γιατί μπόρεσε να ολοκληρώσει την προσπάθεια αυτή για να καταλήξουμε στην συμβιβαστική αυτή λύση και θα είναι πολύ δύσκολο να απομακρυνθεί κανείς από τη λύση η οποία προτείνεται από το Συμβούλιο. Ευχαριστώ. Τώρα είναι μια καλή ευκαιρία οι εισηγητές να δώσουν κάποιες απαντήσεις. Εγώ και ο Λαμασού θα κλείσουμε τη συζήτηση αργότερα, οπότε θα ζητήσω στους άλλους να πάρουν το λόγο. Ο Αλά πρώτος. Θα ήθελα σε ένα σημείο κυρίως να επιμείνω, λέει ο κύριος Λαμασούρ. Ο κύριος Εύκοβιτς και ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου το τόνισαν άλλωστε και έδωσαν και γενικότερα πολλές απαντήσεις και τους ευχαριστώ γι' αυτό. Θα ήθελα εδώ να ευχαριστήσω όλους τους συμμετέχοντες για τις παρατηρήσεις τους, τις κριτικές τους, ιδιαίτερα τα μέλη των κοινοβουλίων των κρατών μελών και να επιμείνω σε αυτό το ο οποίος θα είναι ο ρόλος τους από εδώ και πέρα. Θα πρέπει νομίζω να συνειδητοποιήσουμε όλοι μετά από τη συζήτηση αυτό διαφάνει ότι τη στιγμή κατά την οποία θα συμφωνήσουμε για τον κανονισμό τα τρία θεσμικά όργανα μέχρι το τέλος του χρόνου γιατί αυτό είναι ο πολιτικός στόχος και γυτνιάζουν επαρκώς οι θέσεις μας έτσι ώστε για να μπορέσουμε πράγματι να θεωρήσουμε ότι ο στόχος αυτός είναι ρεαλιστικός. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι πρώτες πρωτοβουλίες θα ξεκινήσουν ήδη από την 1η Ιανουαρίου του 2011. Όχι. Όχι γιατί θα απαιτηθεί ένα εφαρμοστικό εθνικό δίκαιο του ευρωπαϊκού κανονισμού. Στην ουσία έχουμε να κάνουμε κάτι αντίστοιχο με την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Υπάρχουν ευρωπαϊκοί κανόνες οι οποίοι επιβάλλονται σε κάθε χώρα μέλος, σε κάθε κράτος μέλος, αλλά κάθε χώρα έχει επίσης και τους δικούς της εθνικούς, ε, τις δικές της εθνικές ρυθμίσεις. Θα υπάρξουν κάποιοι κοινοί κανόνες για όλα τα κράτη-μέλη, αλλά στη συνέχεια και σχετικά με τον έλεγχο των υπογραφών, αυτός θα εξαρτηθεί εν πολλής από τις εθνικές νομοθετικές ρυθμίσεις. Αυτό θα εξαρτηθεί και από το περιεχόμενο αυτών των κανόνων, αλλά θα εξαρτηθεί επίσης και από τις επιμέρους ρυθμίσεις. Οι εφαρμοστικές αυτές διατάξεις είτε μπορεί να υιοθετηθούν από το εκτελεστικό τμήμα, μέσω ενός διατάγματος σαν παράδειγμα, στη Γαλλία παράδειγμα, αλλά στις περισσότερες άλλες χώρες, ίσως πραγματικά στις περισσότερες, θα πρέπει να χρειαστούν ειδικέ εφαρμοστικές νομικές ρυθμίσεις. Εδώ λοιπόν τίθεται εκ νέου ο ρόλος των Εθνικών Κοινοβουλίων και η παρέμβασή τους θα πρέπει να είναι ταχυτάτη και ιδιαίτερως αποτελεσματική. Τα κοινοβούλια των κρατών μελών λοιπόν θα συμμετάσχουν πλήρως στην επεξεργασία του συστήματος. Δεύτερος ρόλος, τον οποίο καλούνται εφόσον το επιθυμούν να παίξουν τα εθνικά κοινοβούλια, εδώ έχουμε να κάνουμε μια όχι νομική αλλά πολιτική διάσταση, είναι ότι πρόκειται για την παρακολούθηση από κοντά των διαδικασιών αυτών. Διαδικασίες οι οποίες είτε θα επιτύχουν είτε και μπορεί και να αποτύχουν. Αλλά παρόλα αυτά θα έχουν συλλέξει ένα πολύ μεγάλο αριθμό υπογραφών που θα εκφράζουν εν πάση περιπτώσει μια ανησυχία των πολιτών. Και ναι μεν εδώ νομικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα είναι υποχρεωμένη να δώσει συνέχεια, αλλά θα ήταν λάθος πολιτικά να τις αγνοήσουμε τις πρωτοβουλίες αυτές. Αυτό είναι ένα θέμα πάνω στο οποίο θα πρέπει να σκεφτούμε από κοινού ανεξαρτήτως του περιεχομένου του κανονισμού. Έχουμε κάθε συμφέρον να συνεχίσουμε την ανταλλαγή ιδεών εδώ. Διότι η εμπειρία θα δείξει ότι θα υπάρξουν πολλές πρωτοβουλίες οι οποίες θα επισυμβούν σε τομείς οι οποίες είναι κοινή αρμοδιότητας Ευρωπαϊκής Ένωσης και κράτους μέλους. Και για να υπάρξει ικανοποίηση στον πολίτη που συμμετέχει στην διαδικασία αυτή, στην πρωτοβουλία αυτή και εφόσον υπάρχει δηλαδή μια προσδοκία η οποία χρήζει μια απάντηση, θα πρέπει να υπάρξει ένα στοιχείο απάντηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα το προτείνει, η δική της είναι η ευθύνη, και ταυτόχρονα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο φυσικά και το Συμβούλιο Υπουργών. Αλλά θα πρέπει να υπάρξουν στοιχεία απάντησης και σε επίπεδο εθνικής κυβέρνησης, κυβέρνησης κράτους μέλους. Θα πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να μείνουμε σε επαφή έτσι ώστε να μπορέσουμε να δούμε πώς θα χρησιμοποιήσουμε τη διαδικασία αυτή προς το συμφέρον των συμπολιτών μας. Ευχαριστώ. Αλλά... Η Νταϊάννα. Πολλά υπόθηκαν σήμερα το απόγευμα και ήταν ε, για όλους τους συζητητές πολύ χρήσιμα. Ένα σημείο θέλω να θίξω εγώ. Ως αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Γιατί ακούστηκαν πολλά σχόλια που πάνε προς την κατεύθυνση την εξή. ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή άλλα κοινοβούλια αποδυναμώνονται από αυτή τη διαδικασία. Και θα έρθω σε αυτό που είπε και ο Επίτροπος στην αρχή. Το αποτέλεσμα της συνθήκης της Λισαβόνας είναι νικητές από τη διαδικασία να είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα Εθνικά Κοινοβούλια και οι Ευρωπαίοι πολίτες. Να τα τρία στοιχεία που κερδίζουν από τη συνθήκη της Λισαβόνας. Πρέπει λοιπόν να το λάβουμε υπόψη μας αυτό και να συνεργαστούμε μεταξύ μα. Εγώ χαίρομαι που συμμετείχα στις συζητήσεις όπως και ο Επίτροπος για τη συνεργασία των θεσμικών οργάνων στο μέλλον. Όντως έχει ενισχυθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει μεγαλύτερη εξουσία πρωτοβουλίας, έχει συγκεκριμένους τρόπους με τους οποίους καλείται να αντιδράσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αυτό πρέπει να φανεί και στην πρωτοβουλία Ευρωπαίων πολιτών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για παράδειγμα, μπορεί σε τρεις μήνες να φροντίσει να δοθεί απάντηση στους Ευρωπαίους πολίτες. Επίσης, το Κοινοβούλιο θα ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσα σε ένα χρόνο να κάνει μια πρόταση. Και αν δεν το κάνει, θα πρέπει να μας πει γιατί. Το ίδιο θα πρέπει να πει και στους πολίτες. Τα είπανε και ο Αλάν και άλλοι. Αν δεν δοθεί συνέχεια, το πολιτικό κίνημα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και σε εθνικό επίπεδο θα είναι τέτοιο που τα πράγματα θα προχωρήσουν έτσι κι αλλιώς, δεν θα χαθούν. Από μας εξαρτάται να συνεργαστούμε καλά μεταξύ μας. Η ιδέα πάντως ότι το Κοινοβούλιο αποδυναμώνεται με τις ιδέες αυτές είναι κάτι που δεν δέχομαι. Είμαστε όλοι και το Κοινοβούλιο και οι Ευρωπαίοι πολίτες σε καλύτερη θέση τώρα. Ευχαριστούμε. Εσείς ε, σίγουρα, μάλλον από εσά έχουμε να μάθουμε εμείς για το πώς να προεδρεύσουμε μια συνεδρίαση. Προσπαθώ και εγώ να μάθω από εσά. Ο κύριος Έφνερ τώρα έχει το λόγο. Θα ήθελα και εγώ να μιλήσω στη μητρική μου γλώσσα, γιατί σχεδόν όλοι χρησιμοποίησαν τη μητρική τους γλώσσα. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτές τις πολύ ενδιαφέρουσες παρεμβάσεις. Νομίζω ότι θα ήταν πάρα πολύ να τοποθετηθώ σε όλες αυτές λεπτομερώς. Αρκετά ήδη ελέγχθησαν, αλλά πάλι θα τα σκεφτούμε στις πατρίδες μας. Ε, για μένα υπάρχουν ορισμένα πράγματα που είναι σημαντικά. Ε, το ένα είναι ότι θέλουμε ένα εργαλείο για τον πολίτη. Τίποτα άλλο. Γιατί κάποιο είπε ε, να έχουμε ευρωπαϊκές εταιρείε ε, μετά από πρωτοβουλία των πολιτών. Κοιτάξτε, αν ρίξει κανείς ε, μια ματιά ε, στο τι έχει γράψει η Κομισιόν και σε αυτά που λέμε εμείς, δεν πρόκειται για νομικά πρόσωπα. Εμάς μας ενδιαφέρουν τα εργαλεία για τον πολίτη. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι προφανώς και η νομολογία θα πρέπει να αφορά την ουσία των διαδικασιών. Η Κομισιόν προφανώ ανά πάσα ώρα και στιγμή παραμένει ελεύθερη στην αποφασή τη κατά πόσο επιθυμεί να αναλάβει την πρωτοβουλία ή όχι. Εμεί εκείνο το οποίο επιθυμούμε είναι μόνο να υπάρχει μία ε, διαδικασία όπου όσοι αναλαμβάνουν την πρωτοβουλία να νιώθουν ότι αξίζει τον κόπο και όχι ότι αυτά που θα πούνε θα καταλήξουν στον κάλαθο των αχρήστων. Και γι' αυτό το σκοπό συνεργαζόμαστε όλοι. Το τρίτο που θέλω να πω, και με αυτό θα κλείσω, είναι το εξή. Μάλλον, πριν κλείσω. Το παραδεκτό, να το ελέγχουμε στην αρχή, αλλά και παράλληλα να απελευθερώσουμε την Κομισιόν από την πίεση όλα τα νομικά θέματα να πρέπει να τα έχει ε, απαντήσει καταληκτικά εκείνο που οφείλουμε να γνωρίζουμε είναι ότι ε, πράγματι η Κομισιόν έχει το δικαίωμα να καταθέσει πρόταση. Αυτό ε, όμως δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να εξετάσουμε το κατά πόσον δεν γίνεται κατάχρηση όχι. Εφόσον απαντηθούν σε αυτά, τα βασικά θέματα, ε, μετά μπορεί να ακολουθήσει η πρωτοβουλία των πολιτών και η τελική απόφαση σχετικά με το παραδεκτό όχι λαμβάνεται στο τέλος. Άκουσα τις απόψεις όλων. Γνωρίζουμε και τις ε, τοποθετήσεις των κυβερνήσεών σας και οφείλω να επισημάνω ότι υπάρχουν κάποιες ε, διαφορές. Βεβαίως και όλα αυτά σχετίζονται με το τι ρωτάει κανείς και σε ποιον απευθύνεται. Παραδείγματος χάρη, οι κυβερνήσεις ερωτήθηκαν ποια ε, έγγραφα χρησιμοποιούν για να ελέγξουν την ταυτότητα όσων έχουν υπογράψει. Και τους αναφέρθηκε ότι θέλουμε την ταυτότητα, το διαβατήριο, ε, την άδεια κυνηγιού, το ποινικό μητρό και οτιδήποτε. Εμείς αυτή τη στιγμή ρωτάμε περισσότερο τι ακριβώς γίνεται σε διάφορες ε, διαδικασίες όπως συμμετέχουν οι πολίτες. Τι ελέγχεται εκεί. Κατά κανόνα όλα αυτά τα έγγραφα δεν είναι απαραίτητα. Δεν είναι απαραίτητα αυτά που θέλει τώρα η Κομισιόν να χρησιμοποιήσει για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών. Βεβαίω, ε, σε κάποια κρατημέλη υπάρχουν πρωτοβουλίες πολιτών και εκεί αρκεί το όνομα και η διεύθυνση. Αυτό είναι ένα θέμα που θέλουμε να το συζητήσουμε περαιτέρω. Γιατί τελικά εμάς δεν θα μας άρεσε να έχουμε ένα εργαλείο για τον πολίτη το οποίο σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι πολύ πιο γραφειοκρατικό από ότι σε εθνικό επίπεδο. Και αυτό Απλά και μόνο διότι το ζητάνε τα κράτη-μέλη. Και ξέρετε γιατί. Αυτό θα σήμαινε προκαταλήψει απέναντι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή που δεν ε, βασίζονται πουθενά. Παρακαλώ λοιπόν να συζητήσετε με τις κυβερνήσεις σας. Τώρα στο Συμβούλιο θα έχουμε την ε, τελική τριμερή συζήτηση. Εσείς να συζητήσετε με τις κυβερνήσεις για να δείτε κατά πόσο όλα αυτά τα θέματα δεν μπορούν να πληθούν πιο φιλικά προς τον ε, πολίτη και περισσότερο ρεαλιστικά. Είμαστε τυχεροί που έχουμε την πρόεδρο της Επιτροπής Αναφορών μεταξύ μας. Eh, Σε ευχαριστώ που μου δώσατε το λόγο, κυρία Τσίτα Γκουρμάη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον πρόεδρο Καζίνη γιατί συνεννοήθηκε και με τη δική μου επιτροπή την διαδικαστία την οποία θα ακολουθήσουν οι δύο κοινοβουλευτικές επιτροπές. Ε, βρήκα την συζήτηση ιδιαίτερως ενδιαφέρουσα. Είναι μια πρωτοβουλία την οποία προωθήσαμε και εμείς μέσω της Επιτροπής ε, Αναφορών. Το ότι συνεργαζόμαστε με αυτήν εδώ την Επιτροπή είναι κάτι το οποίο διευρύνει θα έλεγα την ειδική μας χαρακτηριστική αρμοδιότητα σε αυτή τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή μου έκαναν θετική εντύπωση και οι παρεμβάσει των εκπροσώπων των κοινοβουλίων των κρατών μελών. Οι περισσότεροι συμφώνησαν και κατανόησαν ορθά κατά τη γνώμη μου τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία σχετικά με αυτό το νέο δικαίωμα το οποίο αναγνωρίζεται. Άκουσα επίσης και σημείωσα μια γενικότερη σύγκληση όχι μόνο ανάμεσα στους εκπροσώπους των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων αλλά και τους εκπροσώπους των κοινοβουλίων των κρατών μελών. Προφανώς και υπάρχουν κάποιες διαφοροποιήσεις. Οι διαφοροποιήσεις αυτές θεωρώ ότι είναι θεμητές εκφράσεις ανησυχιών, αλλά σε καμία περίπτωση διαφοροποιήσεις επί της ουσίας πολιτικού χαρακτήρα. Νομίζω ότι όλοι προσπαθούμε να ανταποκριθούμε με τον πιο πλήρη τρόπο στην μεγάλη ανάγκη η οποία υπάρχει να δώσουμε σάρκα και οστά στο συγκεκριμένο δικαίωμα του πολίτη να συμμετέχει στη ζωή των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να μπορέσει να λειτουργήσει ο πολίτης, με συγχωρείτε για τη φράση που θα χρησιμοποιήσω λίγο υπερβολική, αλλά να συμμετέχει ο πολίτης σαν συνομοθέτης. Ακούστηκαν όμως όπως είπα αρκετές ανησυχίες με κάποιες από αυτές νομίζω ότι και εγώ θα συμφωνήσω. Σαν παράδειγμα για το χρονοδιάγραμμα είμαι υποχρεωμένη να σταθώ λίγο στο χρονοδιάγραμμα. Θεωρώ ότι ε, ακούστηκε από τους περισσότερους ε, η ανάγκη να επιταχυνθούν οι διαδικασίες ολοκλήρωσης της συγκεκριμένης διαδικασίας γιατί οι πολίτες περιμένουν εδώ και αρκετό καιρό και είναι πάρα πολύ δύσκολο να τους εξηγήσει κανείς το γιατί αυτής της χρονικής υστέρησης. Το χρονοδιάγραμμα το οποίο αυτή τη στιγμή προτείνουν οι εισηγητές είναι κάτι το δύσκολο ιδιαίτερα για αυτούς. Αλλά βλέποντας συνολικά το πώς έχουν τώρα τα πράγματα και μετά από τις συζητήσεις διαπραγματεύσεις και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με το Συμβούλιο Νομίζω ότι το χρονοδιάγραμμα μπορεί να τύχει βασμό. Είμαι εξάλλου πεπισμένη λέγοντας ότι τα δύο βασικά έγγραφα τα οποία επεξεργάστηκαν οι συγγητές της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Αναφορών είναι μεταξύ τους εναρμονισμένες εισηγήσεις. Κάποιες διαφοροποιήσεις υπάρχουν, αλλά σχετικά μάλιστα με τον ρόλο της Επιτροπής Αναφορών στην διαδικασία, αλλά νομίζω ότι το αίσθημα ευθύνη όλων θα μας οδηγήσει στην, στο να ξεπεράσουμε τις διαφωνίες αυτές. Θα ήθελα να επανέλθω σε κάποια συγκεκριμένα σημεία, τα οποία παραμένουν ανοιχτά θα έλεγα και τα οποία κυρίως αφορούν στο πρόβλημα του αποδεκτού των συγκεκριμένων πρωτοβουλειών. Εδώ στάθηκαν πάρα πολλοί συνάδελφοι. Είναι σαφές και θα συμφωνήσω με αυτούς ότι θα πρέπει να υπάρξει ε, ένα, μια απλή διαδικασία αλλά ταυτόχρονα τα κριτήρια περί του αποδεκτού ημί και επιμένω σε αυτό, τα κριτήρια λοιπόν θα πρέπει να καθοριστούν με τον πιο συγκεκριμένο δυνατό τρόπο για να, να περιορίσουμε όσο μπορούμε περισσότερο τις αρνητικές απαντήσεις. Και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας την πρόταση την οποία έκανε η κυρία Γκρινή, να συνδέσουμε δηλαδή ήδη από αυτή τη φάση, στη φάση δηλαδή του ελέγχου του αποδεκτού ή μη μιας τέτοιας πρωτοβουλίας και την δυνατότητα αξιολόγησης της πρότασης με έναν αριθμό χαμηλότερο από αυτόν που ε, έχει ήδη προταθεί. Όταν ξεκινάει λοιπόν η διαδικασία συλλογής που θα πρέπει να οδηγήσει στο 1 εκατομμύριο, να ξεκινάει ο έλεγχος μόνο εφόσον έχει ε, γίνει δεκτή ε, η διαδικασία σαν αποδεκτή. Και αυτό θα μας οδηγήσει στο να αποφύγουμε ένα χάσιμο χρόνο και για τον πολίτη και για τα θεσμικά όργανα. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό που είπε η Γκρινή είναι ένα θετικό σημείο, πρέπει να σταθούμε σε αυτό και καλό θα είναι να προσπαθήσουμε να εκτιμήσουμε και τι ρόλο εδώ μπορεί να παίξει η Επιτροπή Αναφορών. Το δεύτερο θέμα και τελευταίο που αφορά τη συνέχεια η οποία θα δοθεί είναι κάτι το οποίο έχει απασχολήσει πάρα πολλούς από αυτούς που πήραν το λόγο Πώς θα πρέπει δηλαδή να συμπεριφερθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέναντι σε μια πρωτοβουλία η οποία έχει ολοκληρώσει την πορεία της, έχει κηρυχθεί αποδεχθεί, αποδεκτή συγγνώμη, και ε, αξιολογείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την μελετά εν σιωπή ή ε, ξεκινάει μια ανοιχτή συζήτηση μέσα από μια ανοιχτή ακρόαση. Αυτό θα το κάνει μόνη της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή θα χρησιμοποιήσει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε εισαγωγικά το χρησιμοποιήσει. και με την Επιτροπή Αναφορών στα πλαίσια του παραδοσιακού ρόλου που έχει η Επιτροπή Αναφορών ως κύριου συνομιλητή του πολίτη. Λοιπόν, νομίζω ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε εδώ να δούμε ποια θα είναι η συνέχεια που θα δίδει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να προσπαθήσουμε επίσης να αξιολογήσουμε με τον πιο συγκεκριμένο τρόπο τα στοιχεία τα οποία θα μπορέσουν να στηρίξουν και να καταστήσουν εφικτή την δυνατότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είτε να εκφράσει μια αρνητική άποψη ή και να δικαιολογήσει ως μη αποδεκτή μια συγκεκριμένη τέτοια διαδικασία. Πάντα σε σχέση με το λεγόμενο follow-up, τέθηκε και το θέμα της επικάλυψης της διαδικασίας αυτής με την διαδικασία αναφορών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Αρμόδια Επιτροπή. Και είπαν ότι σε αυτή την περίπτωση αν δεν γίνει αποδεκτή μια τέτοια λαϊκή πρωτοβουλία ε, να ε, ταξινομηθεί προς τα κάτω αν θέλετε στο επίπεδο των αναφορών, να θεωρηθεί σαν αναφορά. Αυτό νομίζω ότι είναι ένα βήμα το οποίο δεν θα πρέπει να κάνουμε. Θα πρέπει να μην το κάνουμε για να αποφύγουμε μορφές συγχύσεως οι οποίες θα αποδυναμώσουν και θα καταστήσουν την εμβέλεια του συγκεκριμένου αυτού μέσου ιδιαιτέρως περιορισμένη. Οι αναφορές είναι ένα σημείο, αν θέλετε, συναλλαγή σε εισαγωγικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τους πολίτες για να μπορέσουν οι πολίτες να καταγγείλουν πιθανές παραβιάσεις του κοινοτικού νόμου ή κάποιες ασύμβατες ενέργειες των κρατών μελών. Αντίθετα, η λαϊκή πρωτοβουλία είναι μια νομοθετική πρωτοβουλία. Είναι μια δράση η οποία επαφίεται στην πρωτοβουλία των ιδίων των πολιτών έτσι ώστε να μπορέσουν να συνεισφέρουν στην ομοθετική αρμοδιότητα και δραστηριότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κάτι το εντελώς διαφορετικό από αυτά τα οποία αντιμετωπίζουμε εμείς στην Επιτροπή Αναφορών. Συνεπώς έχει σημασία σε όλα αυτά τα σημεία να σκεφτούμε ακριβώς τι θα κάνουμε. Πέραν αυτών θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για την προσπάθεια την οποία κάνατε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω κυρίως τους εισηγητές οι οποίοι μπόρεσαν να καταστήσουν αυτήν την ομάδα συνεκτική και λειτουργική στην αρχή είχαν υπάρξει αμφιβολίες για την εγκυρότητα, αν θέλετε, μια τέτοια θα έλεγα μεγάλη ομάδα εισηγητών. Μετά από αυτούς τους πρώτους μήνες εργασίας όμως μπορούμε να πούμε ότι η επιλογή του να δημιουργηθεί μια μεγάλη ομάδα ήταν μια σωστή επιλογή γιατί η δουλειά που ε, παρήγαγε ήταν εξαιρετική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 Από τη συζήτηση προέκυψαν δύο συμπεράσματα. Ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτή η διαδικασία, κυρίως αυτή η διαδικασία, είναι ψευδεπίγραφη. Εγώ διαφωνώ, διότι θεωρώ ότι ε, το νέο εργαλείο δεν μπορεί να είναι αντικείμενο κατάχρησης θα μπορούσε μάλιστα να εξελιχθεί στο πλέον δημοκρατικό εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι περισσότεροι ε, θεωρούν ότι πρέπει να είναι φιλικό προς τον χρήστη, ε, θεωρούν ότι πρέπει να υπάρχει προστασία δεδομένων. Ε, πρέπει να αποφύγουμε οποιαδήποτε μορφή κατάχρησης. Και θα μιλήσω τώρα αγγλικά. Θέλουμε... Θέλουμε οι Ευρωπαίοι πολίτες να εκμεταλλευτούν αυτή τη νέα πρωτοβουλία και όπως γνωρίζετε όλοι σας αυτή η πρωτοβουλία του πολίτη το να γίνει μια λειτουργούσα πραγματικότητα αυτό χρειάζεται κάποιο χρόνο γι' αυτό λοιπόν είμαι πεπισμένη ότι ε, η Κομισιόν, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πρέπει να αποδείξουν ότι είναι σε θέση να συνεργαστούν. Από δικής μας πλευράς πρέπει να πω ότι δουλεύουμε σκληρά για να υπάρχει το εργαλείο το συντομότερο δυνατόν. Εναπόκειται στα εθνικά κοινοβούλια και στις κυβερνήσεις να δείξουν πόσο γρήγοροι και αποτελεσματικοί είμαστε. Θα ήθελα να σας ζητήσω να έρθετε σε επαφή με τις κυβερνήσεις σας για να ε, γίνουν όλα αυτά πραγματικότητα. Σήμερα λοιπόν πολλά εξαρτώνται από τα εθνικά κοινοβούλια. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι το κοινοβούλιο και η Κομισιόν έχουν δουλέψει πολύ καλά Είμαστε πρόθυμοι να συνεργαστούμε με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Εσείς όμως είστε η φωνή των Εθνικών Κοινοβουλίων. Ε, χρειαζόμαστε λοιπόν τη δική σας τη γνώμη. Θέλω να ευχαριστήσω όλους ε, όσοι παρέμειναν εδώ. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους συναδέλφους από τα Εθνικά Κοινοβούλια, ε, ιδιαίτερες ευχαριστίες προς τους διερμηνείς, ε, στη γραμματεία που ασχολείται με τις σχέσεις με τα Εθνικά Κοινοβούλια, γιατί είναι πολύ δύσκολο να φέρει κανείς εδώ μέλη από 27 κράτη Επίσης ε, η Επιτροπή Αναφορών και η δική μας Επιτροπή ε, αποδείχθηκε ότι μπορούν να συνεργαστούν θαυμάσια και χαίρομαι ε, πάρα πολύ που είμαστε εδώ τρεις γυναίκες στο πόντιουμ αλλά δεν και τυχαίο είχαμε κρίση και αναγκάστηκαν οι άνδρες να παραδώσουν τα ενία σε εμά για να λύσουμε την κρίση τέλος πάντων χαριτολογώντας το από αυτό το θέμα είναι να δούμε πώς θα τα κάνουμε όλα αυτά πραγματικότητα και πώς οι Ευρωπαίοι πολίτες ε, θα ε, ενστερνιστούν τη δημοκρατία. Και ε, στον κύριο Νίτρα θα ήθελα να πω ότι τον παρακαλώ να δείξει στη Σλοβακία ότι πραγματικά μπορούμε να τα καταφέρουμε. Σας ευχαριστώ.